Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir nehmen unsere Beratungen wieder auf mit Tagesordnungspunkt 58. Ξαναρχίζουμε. Η μερίσια διάταξη, σημείο 58, απαλλαγή του Κοινοβουλίου. Ο κύριος Ντένις Δε Γιόγκ έχει το λόγο για να παρουσιάσει την έκθεση. Ορίστε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος. Θα προσπαθήσω τουλάχιστον. Η έκθεση είναι μακρά, αλλά δεν θα επισέλθω σε όλα τα σημεία. Βέβαια, είμαι στη διάθεσή σας για τυχόν ερωτήσεις. Καταρχήν, είναι σημαντικό να αναφερθούμε στην αρχή της έκθεσης, όπου εξέτασα τη συνολική διαδικασία σχετικά με το δημοσιονομικό έλεγχο και το κοινοβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο θεωρεί ότι εδώ πρόκειται κυρίως για δαπάνες προσωπικού και είναι πολύ ε, χαμηλότερο το ποσοστό ε, παρατυπιών. Λίγες συναλλαγές ελέγχθηκαν από το ελεγκτικό συνέδριο. Εγώ μίλησα με κάποιον εκπρόσωπο του συνεδρίου. Το ποσοστό σφάλματος είναι χαμηλό αλλά αν υπάρχουν σφάλματα, αυτό είναι κίνδυνος σημαντικός για το κύρος του Κοινοβουλίου και το βλέπουμε αυτό σε τακτική βάση. Γιατί συχνά βλέπουμε στα μέσα άρθρα και αναφορές σχετικά με το Κοινοβούλιο. Οπότε πιστεύω ότι ίσως πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο στο ζήτημα αυτό και ιδιαίτερα να, βλέπω, να βλέπει το ελεγκτικό συνέδριο και ο προπολογισμό βάσει αποτελεσμάτων. Θα επανέλθω σε αυτό. Αν δούμε επίσης την τεκμηρίωση και τους λογαριασμούς, τα μέλη της Επιτροπής μας θεωρείται ότι είναι ειδικοί στην αξιολόγηση και αποτίμηση των λογαριασμών. Έχουμε πείρα βέβαια σε αυτόν τον τομέα και μπορούμε να βγάλουμε και κάποια συμπεράσματα, αλλά αν το συγκρίνω αυτό με το πώς γίνεται στο Ολλανδικό Κοινοβούλιο, για παράδειγμα, εκεί πριν αρχίσει κανείς την πολιτική αξιολόγηση, κάνει αξιολόγηση των λογαριασμών και του τι περιέχουν. Και οτιδήποτε είναι περίεργο, και αυτό μάλιστα ε, ετοιμάζεται από γραμματεία που έχει, έχει πραγματογνωμοσύνη στην ανάλυση των λογαριασμών και την αποτίμησή τους. Νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε και εμείς κάτι τέτοιο στο Κοινοβούλιο. Δεν χρειάζεται να διευρύνουμε τη Γενική Διεύθυνση ή να χρησιμοποιήσουμε πόρους ε, ε της ΥΠΟ Μπορεί δηλαδή να βρούμε υποστήριξη. Κάποια πραγματογνωμοσύνη χρειάζεται όμως στο μέλλον για να βλέπουμε τους λογαριασμούς. Και αυτό σημαίνει ότι οι έλεγχοι μας θα είναι πιο εξειδικευμένοι. 1,2 δις ε, ε, ευρώ είναι στον προϋπολογισμό μας και αυτό θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Δεύτερον, ε, ασπάθηση, αυτό θα πρέπει να το δούμε σε σχέση με τον προϋπολογισμό βάση επιδόσεων. Έχει γίνει εξαιρετική δουλειά στο Κοινοβούλιο και έχω γράψει κάποιες σχετικές παραγράφους. Και ορισμένα, σε ορισμένα σημεία το Κοινοβούλιο έχει πολύ ε, συγκεκριμένη προσέγγιση, αλλά με απασχολούν η πολιτική των επικοινωνιών. Έχει συζητηθεί πολύ το θέμα και στο παρελθόν, δηλαδή το βραβείο Λουξ. και το Ευρωπαϊκό Σπίτι της Ιστορίας, Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας, γραφεία ενημέρωσης επίσης και θα και ζητώ στο σχέδιο έκθεσης το ελεγκτικό συνέδριο να εξετάσει συγκεκριμένα την πολιτική επικοινωνιών όχι μόνο του Κοινοβουλίου αλλά ευρύτερα και να δει πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τον προϋπολογισμό βάσει επιδόσεων σε αυτό το τομέα και πώς μπορούμε να φτάσουμε το μήνυμά μας σε ανθρώπους που δεν δείχνουν αυθόρμητα ενδιαφέρον για τα ευρωπα... τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Αυτό είναι μια πρόκληση για τους πολιτικούς γενικότερα, γιατί βλέπετε μια γενικότερη δυσαρέσκεια σήμερα ε, απέναντι στην πολιτική και θα πρέπει να δούμε πώς θα έρθουμε σε επαφή με αυτούς τους ανθρώπους, πώς να τους αγγίξουμε. Ε, εκεί δεν έχω δει ιδιαίτερα καινοτόμε ιδέες. Παλιά αποστέλναμε κάποια μηνύματα, αλλά δεν ακούγαμε. Δεν υπήρχε διάδραση. Επίσης, το, ευρωπαϊκό, το σπίτι της ευρωπαϊκής ε, ιστορίας είναι δουλειά του Κοινοβουλίου. Πρέπει να το δούμε και αυτό, το σπίτι της ευρωπαϊκής ιστορίας. Ε, ε, αυτό το θέμα γίνεται λίγο σαν τουριστική ατραξιόν στις Βρυξέλλες. Πρέπει να κάνουμε κάτι, να κάνουμε συζητήσεις στις Βρυξέλλες για το πώς θα γίνει και ο γειτονικό χώρος πιο ελκυστικός ως αποτέλεσμα αυτών των δυνατοτήτων και πώς μπορούμε να συμβάλλουμε με διάφορους τρόπους. Σίγουρα κάτι πρέπει να κάνουμε και εδώ. Ε, η διαφάνεια δαπάνες ταξιδίου, αυτό το ακούμε σε σχέση με το Γενικό Γραμματέα, τα websites, προσωπικά websites, ή ιστοσελίδες δηλαδή του κάθε ευρωβουλευτή και πώς μπορούν να βελτιωθούν και ε, άλλα ε, ζητήματα. Επίσης, το προαιρετικό συνταξιδοτικό ταμείο, ταμείο συντάξεων, ε, που υπήρχε μέχρι το 2009, απειλείται από μεγάλα ελλείμματα στο μέλλον. Οι ε, ε, Ολλανδοί δημοσιογράφοι μου επέστησαν την προσοχή με ερωτήσεις πάνω σε αυτό και στον Ολλανδικό τύπο είναι ένα επανερχόμενο θέμα. Είναι ιδιαίτερα προβληματικό σήμερα γιατί εδώ υπάρχει πολύ χαμηλό ε, ποσοστό κάλυψης, 37%. το σύνηθες, ε, η, σύνηθι, η κάλυψη είναι 105% για ένα τέτοιο ταμείο συντάξεων. Και κάναμε και περικοπές ε, συντάξεων για να κρατήσουμε την αναλογία στην Ολλανδία. Ε, είναι διαφορετική η δομή από ό,τι στις συνήθεις επιχειρήσεις, αλλά εδώ, σε τελευταία ανάλυση, όλα αυτά τα ελλείμματα θα τα πληρώσει ο φορολογούμενος. Άρα πρέπει να βρούμε μια διαφορετική λύση. Ε, κάποιοι πρώην ε, ευρωβουλευτές ε, εξακολουθούν να συμβάλλουν με κάποια μικρά ποσά, ακόμα δεν λαμβάνουν σύνταξη και ίσως θα μπορούσαμε να βρούμε κάποια ρύθμιση και με αυτούς που παίρνουν σύνταξη, ούτω ώστε να μην πληρώνουν τα σπασμένα οι φορολογούμενοι. Το πρόβλημα είναι περίπλοκο γιατί υπάρχουν και κάποιες νομικές υποχρεώσεις, αλλά αυτό είναι ένα θέμα ευάλωτο για μας. Ένα άλλο ευάλωτο ε, όχι μόνο για το Κοινοβούλιο όμως αυτό, είναι ότι οι συντάξεις των Ευρωπαίων αξιωματούχων των υπαλλήλων πληρώνονται από την Κομισιόν, αλλά δεν έχει βρεθεί λύση, για παράδειγμα, στην περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου. Αν δηλαδή αποχωρήσει από την Ένωση ένα κράτος μέλος, τις συντάξεις ποιος θα τις πληρώσει. Η Βρετανική κυβέρνηση εμπροκειμένο. Αλλά οι υπάλληλοι θα είναι στο έλεος της εθνικής κυβέρνησης και της απόφασης που θα λάβει. Ένα άλλο σημαντικό είναι τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα. Ε, είχαμε μια συνάντηση κλειστή πάνω σε αυτό το θέμα όπου εγώ κατέθεσα έναν αριθμό προτάσεων για το πώς μπορούν να βελτιωθούν οι έλεγχοι. Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν, έχει γίνει τίποτα. Υπήρξαν διάφορα σκάνδαλα σχετικά με τα κόμματα, τα πιο πρόσφατα μάλλον παρά τα παλιά και εδρεωμένα. Και έχει αναλυφθεί κάποια δράση. Όμως πολύ συχνά οι δημοσιογράφοι δίνουν πληροφορίες που δεν τις έχουμε λάβει εμείς εσωτερικά. Ο Ένστε Γιόγκ, για παράδειγμα, είχε κάποιες πρόσφατες πληροφορίες. Είναι ένα εσωτερικό πρόβλημα αυτό, αλλά και μια δυνατότητα για το μέλλον. Η αρχή που θα αρχίσει να εργάζεται φέτος έχει περιορισμένο προσωπικό και θα εξαρτάται στην πραγματικότητα από τη διοίκηση που επίσης έχει λίγους ανθρώπους να εργάζονται σε αυτό το τομέα. Πάντως κάτι πάμε να κάνουμε και όταν ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία της απαλλαγής θα έπρεπε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα να συνέλθουν για να δουν τι νέα μορφή συνεργασίας μπορούμε να έχουμε με την αρχή αυτή, την αρμόδια αρχή, για να βελτιώσουμε το δημοσιονομικό έλεγχο και η Επιτροπή Κοντ να μπορεί να κάνει ε, ε, έρευνες με βάση το υλικό που παίρνουμε από τα μέρη και τα κόμματα. Τώρα, μια άλλη πολιτική φύσεως μάλλον παρατήρηση που έχει τεθεί και από την Πρόεδρο επίσης είναι το θέμα των καταχρήσεων και ενδεχομένως νεποτισμού από τον πρώην Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρτιν Σούλτς. Ε, έγιναν συμπληρωματικές ερωτήσεις που κατετέθησαν και είμαι βέβαιος ότι αυτό το θέμα θα ξανά έρθει στην επιφάνεια. Στην περσινή έκθεση, την έκθεση του κυρίου Πίπερ, έχει εξεταστεί το ζήτημα. Τώρα προστίθενται νέες πληροφορίες. Θα είναι όμως δύσκολο να ενσωματωθούν στην έκθεση. Εγώ ως εισηγητής πιστεύω ότι είναι καθήκον μας ως Επιτροπή να δούμε με αντικειμενικό τρόπο τα γεγονότα, τα στοιχεία και να ελέγξουμε σε ποιο βαθμό έχουν καλυφθεί από προηγούμενα ψηφίσματα ή έρευνες. Αν υπάρχουν εκρεμή ζητήματα, σίγουρα μπορούμε στη φετινή έκθεση να προσθέσουμε σχετικές συστάσεις, αλλά άμα είναι επανάληψη των ιδίων, δεν ξέρω αν έχει νόημα, αφού δεν οδηγούμεθα σε πρόσθετες δράσεις και έρευνα. Εγώ αυτό το κριτήριο θα χρησιμοποιούσα. Ε, αυτό που είναι σημαντικό εδώ είναι ότι η πολιτική διορισμών των γενικών διευθυντών στηρίζονται σε συμβουλευτική επιτροπή που λειτουργεί εδώ στο Κοινοβούλιο αλλά σε αυτή την επιτροπή είναι μόνο τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη, γενικοί διευθυντές από κάποιες γενικές διευθύνσεις. Αυτοί απαρτίζουν την επιτροπή. Και αν θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρχουν παρατυπίες, θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και τα μεσαία στελέχη της διοίκησης, να έχουν δηλαδή και εκείνοι μεγαλύτερη εκπροσώπηση στη Συμβουλευτική Επιτροπή, γιατί αυτό το παράπονο ακούμε από τους υπαλλήλου. Δηλαδή ε, αν κάποιος θέλει να σταδιοδρομήσει εδώ θα πρέπει να λάβει υπόψη του και κάποιες πολιτικές ε, που θα πρέπει να ακολουθήσει για να φτάσει στην κορυφή. Πάντως θα πρέπει να πάρουμε μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρχουν παρατυπίες στο μέλλον. Αυτά από την πλευρά μου. Ευχαριστώ και θα απαντήσω και σε ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Όπως κάθε χρόνο δημιουργούνται προβλήματα σε σχέση με την απαλλαγή. Χρόνια ε, συμβαίνει αυτό και βεβαίως όλα αυτά τα φορτώνεται όπως και ο κύριος ε, ε, Ντεγιόν. Τώρα ήρθε η σειρά σας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστήσω και τον εισηγητή μας, τον κύριο Ντεγιόνγκ, για την πλήρη αυτή παρουσίαση που έκανε και γενικά ισορροπημένη παρουσίαση της έκθεσης, του σχεδίου έκθεσης. Συμφωνούμε σε πολλές από τις επικρίσεις που τονίζετε και εσείς στην εκθεσή σας και όντως έχουμε έναν πλήρη κατάλογο στην εκθεσή σας. Για παράδειγμα, έλλειψη αποδοτικότητας της στρατηγικής επικοινωνίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το ότι θα πρέπει το βραβείο Λουξ πραγματικά να ανταποκρίνεται στο κόστος του, να δημιουργεί προστιθέμενη αξία. Το κόστος και η διακυβέρνηση του σπιτιού της ευρωπαϊκής ιστορίας ότι έχουμε όλο και περισσότερο κόστο όσον αφορά το σταξιδωτικό ταμείο. Το ότι θα πρέπει να βελτιωθεί επίση η τεχνολογία που χρησιμοποιεί η διεύθυνση ITEC. Νομίζω όμω ότι θα πρέπει να τονίσουμε και την άλλη πλευρά των πραγμάτων. Δηλαδή το ζήτημα τη διαφάνεια. Προφανώς εμείς δίνουμε μάχη για το ζήτημα αυτό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αλλά δεν είμαι πεπισμένος για το αν πραγματικά ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τη διαφάνεια είναι ο πλέον κατάλληλο, ενδεχομένω εδώ να οι απόψει για το πώ μπορούμε να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί στον τομέα τη διαφάνεια. Στην έκθεση, για παράδειγμα, προτείνεται από εσά ότι όλα τα σχετικά έγγραφα που έχουν να κάνουν με τι δαπάνε θα πρέπει να κοινοποιούνται και θα πρέπει να εμφανίζεται στην ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου κάθε τυχόν τέτοιο έγγραφο το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί, ότι θα πρέπει όλα αυτά τα έγγραφα να καταστούν δημόσια. Εγώ και η πολιτική ομάδα δεν είμαστε πεπισμένοι ότι θα πετύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα μια τέτοια προσέγγιση. Έτσι λοιπόν όσον αφορά το τμήμα αυτό της διαφάνειας, ενδεχομένως εμείς να καταθέσουμε κάποιες τροπολογίες εξ του ΕΛΚΑ. Επίσης, Πολλές από τις ε, πληροφορίες που μας ζητάτε ήδη είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και θα έλεγα ότι η σημαντικότερη ανησυχία που έχουμε έχει να κάνει με την ε, αύξηση του διοικητικού κόστους. Και όχι μόνο το κόστος αυτό καθεαυτό, δεν αναφέρουμε μόνο στο τίμημα το θα μπορούσε να έχει μια τέτοια απέτηση, αλλά ανησυχώ ακόμα περισσότερο για το ότι ενδεχομένως να δημιουργηθεί εδώ πέρα ένα πολύ μεγάλο μπέρδεμα, για να το πω με απόλυτη ειλικρίνεια. Πολύ φοβάμαι ότι ε, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξεκαθαρίσουμε εδώ πέρα τα πράγματα και πάλι δεν αναφέρομαι σε δαπάνε. Φοβάμαι ότι θα δημιουργήσουμε ένα πολύ πολύπλοκο διοικητικό σύστημα αν ακολουθήσουμε ακριβώ κατά γράμμα τι συστάσει του σχεδίου εκθεσή σα. Συνεπώς, στηρίζουμε την διαφάνεια, όπως σας είπα, αλλά ενδεχομένως να πρέπει να εξετάσουμε λίγο περισσότερο το πώς θα πετύχουμε το ευκταίο αυτό επίπεδο διαφάνειας. Όσον αφορά τώρα τις πολιτικές ομάδες και τα ιδρύματα πολιτικών ομάδων. Ο γενικότερος στόχος εδώ πέρα μας βρίσκει σύμφωνος. Το πρόβλημα κατά την άποψή μας έγκυται στο ότι αν δούμε τα πιθανά προβλήματα τα οποία μπορούν να προκύψουν από τη χρησιμοποίηση κονδυλίων ή αυτά που προκύπτουν επί του παρόντος, βλέπουμε ότι υπάρχουν τεράστιες διαφορές ανάμεσα στα διάφορα πολιτικά κόμματα. Αυτό το γνωρίζουμε όλοι μας, έτσι δεν είναι. Αν πάρουμε κάθε πολιτική ομάδα ή κάθε πολιτικό κόμμα ξεχωριστά, συνειδητοποιούμε ότι υπάρχουν τεράστιες αποκλήσεις. Για παράδειγμα, γνωρίζω εγώ ότι θα πρέπει να ακολουθήσω συγκεκριμένες προποθέσεις προκειμένου να ακολουθήσω τη γραμμή 400 του προπολογισμού. Τι δικαιολογητικά θα πρέπει να καταβάλω προκειμένου να πάω στη Λαπωνία, για παράδειγμα. Και στη συνέχεια πρέπει να καταβάλω συγκεκριμένα δικαιολογητικά, να πω ακριβώς πώς συμμετείχαν στη συνεδρίαση και το καθεξής. Είμαι υπέρ των αυστηρών αυτών ελέγχων, αλλά τα κριτήρια αυτά ήδη υπάρχουν. Οι προποθέσει αυτές ήδη υφίστανται. Και αν απευθυνθείτε στη διοίκηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα συνειδητοποιήσετε ότι οι κανόνες αυτοί ήδη υφίστανται και ουσιαστικά είναι η μέγιστη δυνατή προκειμένου να επιτευχθεί αυτή η διαφάνεια. Δεν νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να πάμε πολύ καλύτερα. Του λεχθέντων θα καταθέσουμε μια σειρά τροπολογιών για τα ζητήματα αυτά τα οποία έθιξα. Και για άλλη μια φορά, κύριε Σιγητά, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω και είμαι πεπισμένο ότι θα καταφέρουμε να συζητήσουμε περαιτέρω επικοδομητικά όλα αυτά τα ζητήματα στο πλαίσιο της εξαιρετικής σας έκθεσης. Σας ευχαριστούμε κύριε Ντεγιόνγκ, Ολοκληρώνω σε αυτό το σημείο. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφος Γκάιερ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ επικεντρώνομαι στο τελευταίο θέμα που έθιξε ο κύριος Ντε Jong. Νομίζω ότι πολύ σωστά παρουσίασε στο θέμα συνοπτικά. Δηλαδή, ε, αποφάσει για το προσωπικό του πρώην Προέδρου θα πρέπει να δούμε τι είναι καινούριο και τι δεν καλύπτεται στην περσινή έκθεση που δεν με βρήκε σύμφωνο τότε ε, βεβαίως, ως προς τη διαδικασία ε, έχεις δίκιο και έχεις την υποστήριξη πολλών μελών της ομάδας μου. Διότι πρέπει να είναι ξεκάθαρο για μας ως Επιτροπή ότι η έκθεση αυτή και η εργασία αυτή που κάνεις ε, είναι ε, στη δημοσιότητα και θα παίξει ρόλο και στην προεκλογική εκστρατεία στη Γερμανία. Και σίγουρα θα παίξει ρόλο και στο Γερμανικό Κοινοβούλιο. Είναι πολύ σωστό έτσι όπως προχωρείς Τώρα, το ερώτημα είναι υπάρχουν παραβιάσεις κανόνων ή υπάρχουν διαδικασίες που πρέπει να ξεκαθαριστούν, πρέπει να διαλευκανθούν ε, ως προς τους κανόνες που ισχύουν και παρα... δεν ε, εφαρμόστηκαν. Και από τα έγγραφα που έχω και από τη διοίκηση βλέπω αντιφάσεις. Ας πούμε τα υπηρεσιακά ταξίδια. Δεν ξέρω έτσι πως έχουν ρυθμιστεί αν είναι η καλύτερη λύση για το κοινοβούλιο. Γιατί αν είναι η καλύτερη λύση κανένα πρόβλημα. Να συνεχίσουμε. Δηλαδή ε, υπάρχει κάτι ε, για να επικρίνουμε τον Μάρκους Έγγελς ή όχι. Ε, ο, ο, ο ρόλος της Επιτροπής μας δεν είναι απλώς να διαπιστώνει τυχόν παρατυπίες, αλλά να δώσει εναλλακτική και να καλέσει τη διοίκηση να επιλέξει διαδικασίες που θα είναι για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι πλέον οικονομικές. Και παράλληλα θα υπάρχει και ε, σαφήνεια ως προς τους κανόνες και αν αυτοί παραβιάζονται. Είναι δύσκολη η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Υπάρχει η δεδηλωμένη ε, ο δεδηλωμένος ισχυρισμός της διοίκησης ότι δεν υπάρχει πρόβλημα Στη Γερμανία όμως διαβάζω ότι υπάρχει πρόβλημα σχετικά με τους κανόνες. Εδώ πρέπει και η Επιτροπή μας να βρει το ρόλο της. Ε, μπορεί να διαφοροποιηθεί από τη διοίκηση. Εκεί που δεν βλέπει πρόβλημα η διοίκηση, μπορεί η Επιτροπή μας να το δει. Και αυτό θα πρέπει να έχει επιπτώσεις στη διοίκηση. Ευχαριστώ. Περιμένουμε να ε, πάρει θέση η διοίκηση του Κοινοβουλίου. Δεν ξέρουμε ακόμα αν υπάρχει παραβίαση γιατί δεν υπάρχει ε, θέση. Είχαμε πει ότι 3 Μαρτίου θα ε, υπήρχε, ελπίζω έγκαιρα να δοθεί για να μπορούμε να τη μελετήσουμε λεπτομερώς. Ο συνάδελφος ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς να ευχαριστήσω και εγώ τον εισηγητή μας, τον κύριο Ντεγιόγκα, για την εξαιρετική αυτή έκθεση, το εξαιρετικό σχέδιο έκθεσης, το οποίο αποτελεί πολύ θετική βάση για περαιτέρω συζητήσεις. Και όλος ιδιαιτέρως θα ήθελα να χαιρετήσω κάποιες από τις ιδέες που προβάλλονται στην έκθεση, όπως για παράδειγμα το ότι θα πρέπει να υπάρχει υποστήριξη για τα μέλη της Επιτροπής ε, ΚΟΝΤ, ότι θα πρέπει να έχουμε ένα προπολογισμό βάση επιδόσεων, ότι θα πρέπει να υπάρχει μια μοναδική έδρα ή μια πρόθεση, αν θέλετε, στήριξη πρωτοβουλία για μια μοναδική έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θέμα το οποίο έχει ανακύψει πάρα πολλέ φορέ. Και επίση θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει μια πιο εξατομικευμένη στο σελίδα για τους ευρωβουλευτές όπου να παρέχονται περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τις αποζημιώσεις ή όσον αφορά τους εκπροσώπους από τις ομάδες πίεσης με τους οποίους έρχονται σε επαφή οι ευρωβουλευτές. Στον λίγο χρόνο που έχω θα ήθελα να θίξω κάποια ζητήματα από την οποία θεωρώ ότι υπάρχει ένα περιθώριο βελτίωσης. Καταρχάς, τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα σχετικά ιδρύματα και η χρηματοδότησή τους. Υπάρχουν παράγραφοι στην έκθεσή σας γι' αυτό. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι εδώ πέρα θα μπορούσατε να ήσασταν λίγο πιο αυστηρός και σχετικά με τις παραγράφους αυτές θα καταθέσω κάποιες ε, τροπολογίες προκειμένου να έχουμε πιο συστημικούς ελέγχους για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων. Δεύτερον, οι γενικές δαπάνες και αποζημιώσεις γενικών δαπανών Έχουμε κάνει μια εκτενέστατη συζήτηση στο παρελθόν για το ζήτημα αυτό και προφανώ δεν μπορούμε να το επιλύσουμε μόνο στα πλαίσια τη έκθεση αυτή απαλλαγή. Παρ' αυτά θα πρέπει να λέμε ξεκάθαρα ότι πρόκειται για δημόσια κονδύλια και ότι ε, η χρησιμοποίηση των δημόσιων κονδυλίων θα πρέπει να γίνεται με απόλυτη διαφάνεια. Υπάρχουν πολύ διαφορετικοί τρόποι για να εξασφαλίσει κανεί τη διαφάνεια και θεωρώ ότι ε, οι ανησυχίε που ακούστηκαν σε σχέση με την ε, δημοσιοποίηση ακόμα και του κόστους για οποιοδήποτε καφέ πίνει κανείς ή για το οποιοδήποτε ευρώ δαπανά ενδεχομένω να μην είναι προτάσεις ιδιαίτερα ρεαλιστικές θα μπορούσαμε να θέσουμε ένα κατόφλι για παράδειγμα δαπάνες που περβαίνουν τα 100 ευρώ αυτές μόνο να κοινοποιούνται μια ιδέα είναι αυτή ή δεν θα πρέπει να καταλήξουμε σε ένα σύστημα που οι ευρωβουλευτέ αναγκάζονται να δημοσιοποιούν τι αποδείξει του για οποιαδήποτε ακόμα και μηδαμινή δαπάνη ενδεχομένω να έχουν κάνει. Και το ακούσαμε και από τον Προλαλήσαντα ότι ενδεχομένω μπορεί να δημιουργηθεί εδώ πέρα πολύ μεγάλο μπέρδεμα. Ναι, μπορεί να δημιουργηθεί πολιτικό μπέρδεμα, θα έλεγα, γιατί ε, Ξέρω ότι υπάρχουν ορισμένοι συνάδελφοι, ευρωβουλευτέ, οι οποίοι χρησιμοποιούν τον φάκελο αυτό αποζημιώσεων που υφίσταται ω επιπλέον μισθό. Προφανώ λοιπόν αυτό θα πρέπει να αποφευχθεί. Α πετύχουμε λοιπόν την κατάλληλη ισορροπία προκειμένου να υπάρχει αφενό διαφάνεια και από την άλλη χαμηλό διοικητικό άχθο. Πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη μα και το ζήτημα τη ελευθερία των βουλευτών κατά τη διάρκεια τη εντολή του, αλλά και αυτό μπορούμε να το συνδυάσουμε, δηλαδή να έχουμε την απαραίτητη διαφάνεια χωρίς να δημιουργούμε προβλήματα στην εξαρτησία των ευρωβουλευτών. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει προκειμένου να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και ιδίω την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών απέναντι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ένα τρίτο τώρα ζήτημα που θέλω να δείξω, οι εσωτερικοί κανόνε όσον αφορά του καταγγέλτε, του πληροφοριοδότε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει πολύ καλούς κανόνες αυτή τη στιγμή όσον αφορά του καταγγέλτες. Υπάρχουν κάποια προβλήματα ίσονος σημασίας, ιδίως ε, όσον αφορά τα άτομα εκείνα τα πιστοποιημένα, τα οποία συνεργάζονται με τους ευρωβουλευτές και θα πρέπει και αυτά να χαίρουν της κατάλληλης προστασίας. Όσον αφορά τώρα τις παραγράφους που έχουν να κάνουν με το μα. Υπάρχουν κάποια ζητήματα για τα οποία θα ήθελα να καταθέσω τροπολογίες. Δύο επιπλέον σημαντικά ζητήματα. Πρώτον, το ζήτημα των ε, παράλληλων εργασιών που θα μπορούσε να λάβει κανείς. Ε, ξέρετε ότι αυτό το είχαμε θίξει και στην προηγούμενη έκθεση απαλλαγή και είχαμε πει ότι θέλαμε να το διευθετήσουμε το ζήτημα αυτό. Δεν είχαμε όμω τις απαραίτητε ψήφους ε, στην ψηφοφορία που έγινε στην Ολομέλεια και έτσι παράγραφοι από την έκθεση της προηγούμενης χρονιάς ουσιαστικά διαγράφηκαν από την έκθεση. Το ζήτημα όμως υφίσταται και Κάθε φορά που η Επιτροπή μας θέλει να κάνει κάτι με άλλες εργασίες που ενδεχομένω να έχουν ευρωβουλευτές, δυστυχώς δεν έχουμε την απαραίτητη υποστήριξη από τους ευρωβουλευτές. Το πρόβλημα όμως εξακολουθεί να υφίσταται. Και δεύτερον, το ζήτημα που είχε να κάνει με τον Μάρτιν Σούλτς. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να θέσουμε ρητό στα όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του 2014 και Μπορούμε να το κάνουμε αυτό στα πλαίσια, μπορούσαμε να το κάνουμε μάλλον αυτό, στα πλαίσια της προηγούμενης έκθεσης απαλλαγής. Οι πράσινοι μας είχαν υποστηρίξει μέχρι το τέλος της διαδικασίας. Είχαμε πει ότι μαζί τους θέλαμε να θέσουμε κάποια ερωτήματα όσον αφορά τη δραστηριότητα του Μάρτιν Σούλτς, αλλά πάλι φτάσαμε στην Ολομέλεια και εκεί πέρα δεν είχαμε την απαραίτητη υποστήριξη από την πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και για αυτό το ζήτημα. Όπω δηλαδή σκοτώσαμε εντό εισαγωγικών τι παραγράφου εκείνε που είχαν να κάνουν με τι επιπλέον εργασίε που επιτελούν οι Ευρωβουλευτέ, έτσι δεν είχαμε την απαραίτητη πλειοψηφία για να υποστηρίξουμε τι παραγράφου εκείνε που ζητούσαν μια περαιτέρω διερεύνηση όσον αφορά τι δραστηριότητε του Μάρτιν Σούλτ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε πώ έχουν τα πράγματα. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε μια προκλογική εκστρατεία στη Γερμανία. Υπάρχουν λοιπόν κάποιε πολιτικέ ευαισθησίε. Πέρα από αυτό όμω τονίζω ότι από διαδικαστική πλευρά είχαμε στο παρελθόν, συγκεκριμένα πέρυσι, την ευκαιρία να διευθετήσουμε το ζήτημα αυτό και δυστυχώ χάσαμε αυτή την ευκαιρία. Και μου φαίνεται περίεργο αυτή τη στιγμή ότι ανακύπτει εκ νέου το ζήτημα αυτό ω ζήτημα το οποίο πρέπει να επιληθεί, μόνο ότι είχαμε τη δυνατότητα, όπω σα είπα, να το επιλύσουμε πέρυσι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι κύριε Ντεγιόγκ. Θα ήθελα καταρχάς να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την έκθεση που είναι πολύ περιεκτική, ε, παρόλο που είναι περίπλοκο το ζήτημα, είναι πολύ λεπτομερής καλύπτει όλες τις πτυχές ε, της λειτουργίας ε, του Κοινοβουλίου από οικονομικής απόψης είναι πολύ σημαντική ε, όχι μόνο λόγω των πιστώσεων πληρωμών 20% στο πλαίσιο του δημοσιονομικού πλαισίου αλλά και η ορατότητα των δραστηριοτήτων του Κοινοβουλίου είναι πολύ υψηλή και πιστεύω ότι με όλες αυτές τις πτυχές που αναφέρθηκαν θα έπρεπε να είμαστε πολύ προσεκτικοί ε, ποιος θα είναι ο αντίκτυπος στην κοινή γνώμη στην Ευρώπη. Για μας ε, το να προχωρήσουμε παραπέρα δεν ε, έχει να κάνει μόνο με το επίπεδο δαπανών όπως επίσης και με τις παρατυπίες που έχουν εντοπιστεί αλλά και πώς έχουν δαπανηθεί τα ποσά και τι αποτελέσματα έχουν επιτευχθεί με αυτά τα ποσά. Αυτή η προσέγγιση έχει ενσωματωθεί στην έκθεση του κυρίου Ντε και φάνηκε και από αυτά που μας είπε και πιστεύω ότι μια προσέγγιση ε, προϋπολογισμού βάσει δραστηριοτήτων και καλύτερης επίδοσης νομίζω ότι είναι ε, το καλύτερο που μπορούμε να επιθυμούμε. Όσον αφορά το θέμα τώρα της ε, κατάρτισης του προσωπικού και τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί σχετικά για μένα είναι δύσκολο, ε, όπως είπε και ο κύριος Διόγκ, ε, να βρεθούν και άλλες πληροφορίες για τις άλλες πτυχές, πώς μπορεί να προσμετρηθούν αυτά τα αποτελέσματα, δεδομένου ότι έχουν ε, χρησιμοποιηθεί δημόσιοι πόροι για την κατάρτιση. Πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα αξιολόγησης για το πώς υπάρχει προστιθέμενη αξία από την κατάρτιση για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ποσοτικούς όρους. Ευχαριστώ. Συνάδελφε Σμιτ, ευχαριστώ. Όσο πιο πολύ ακούω, τόσο πιο πολύ ενδιαφέρον παίρνει το θέμα. Καταρχήν έχουμε εμπιστοσύνη και στο Κοινοβούλιο και στη Γενική Γραμματεία. Υποθέτω ε, ότι και εγώ είμαι υπέρμαχος της διαφάνειας όπως οι περισσότεροι και γι' αυτό ήταν ενδιαφέρον τις τελευταίες μέρες και εβδομάδες ότι πήραμε στοιχεία, νούμερα από τον τύπο που αφορούν τον πρώην πρόεδρο. Ε, υπάρχουν, υπάρχουν μομφές εναντίον του, οι οποίες πρέπει κατεπηγόντως να διελευκανθούν, όπως είπε και ο συνάδελφος De ε, και παλιά υπήρχαν προβλήματα, αν όμως και τώρα υπάρχουν θέματα, σίγουρα πρέπει να ενσωματωθούν την έκθεση που θα εγκριθεί από την Επιτροπή μας. Θα πρέπει δηλαδή να πούμε και για τις επικρίσεις και να πάρουμε θέση υπέρ του ότι πρέπει να ξεκαθαριστούν όλα τα θέματα. Διότι ότι βρίσκεται γενικώ ε, στον αέρα και εωρείται ως μομφή δεν αφορά μόνο τον Πρόεδρο αλλά και το Κοινοβούλιο. Είναι ένα βάρος αυτό ε, για το Κοινοβούλιο. Δεν ξέρω αν μέχρι 3 Τρίτου ο Γενικός Γραμματέας θα προλάβει να απαντήσει είτε προφορικά είτε γραπτά, πάντως το συντομότερο να υπάρξει ένα δεύτερο follow-up. Νομίζω ότι πρέπει η έκθεση αυτή να λέει τι σημαίνει ε, υπηρεσιακό ταξίδιο μακράς διαρκείας, ποιος μπορεί να κάνει τέτοιο ταξίδι, ποιος αποφασίζει για ένα τέτοιο ταξίδι και ποιος το ελέγχει για να ε, είναι σαφής η νομιμότητα των δαπανών. Ο συνάδελφος Γκάιερ μίλησε για την προεκλογική εκστρατεία. Βεβαίω, είμαστε σε προεκλογική εκστρατεία και στη Γερμανία και τη Γαλλία και την Ολλανδία. Αλλά η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού δεν μπορεί να ε, λαμβάνει τέτοιες παραμέτρους υπόψη της. Ε, παρόλο που μπορεί να υπάρξουν προβλήματα για τον πρώην Πρόεδρο. Είδαμε τα δημοσιεύματα στο Spiegel. Ο κύριος Έγγελς αναφέρεται ως πρώην βοηθός του Προέδρου. Ξέρουμε ότι ήταν πάρα πολύ στις Βρυξε... στο Βερολίνο και όχι στις Βρυξέλλες όπως έπρεπε. Ήταν, λέει, σε μόνιμο υπηρεσιακό ταξίδι Ξέρουμε επίσης ότι έπαιρνε και ημερήσιο επίδομα, αποζημίωση ε, και αποζημίωση επειδή ήταν σε άλλη χώρα, ενώ ζούσε στο Βερολίνο στο σπίτι του. Και δεν ξέρουμε εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέλαβε και να πληρώνει το ενοικιό του. Αυτό είναι μια εσωτερική ρύθμιση. Εγώ θέλω να τα γνωρίζω όμως αυτά. Συνέβη κάτι τέτοιο ή όχι. Επίσης, πήραμε πληροφορίες σχετικά με το πόσα τέτοια διαρκείας υπηρεσιακά ταξίδια ε, γίνονται. Έχουμε στοιχεία από τον τύπο, αλλά πρέπει να τα δίπλο τσεκάρουμε. Θα ήθελα να γνωρίζω στοιχεία σχετικά με το, τα ταξίδια αυτά και ε, ποια τμήματα αφορούν, ποιοι τους έστειλαν και νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε και τη συχνότητα αλλά και τη διάρκεια αυτών των υπηρεσιακών ταξιδίων. Όλα αυτά θα πρέπει να βρεθούν και να μας υποβληθούν. Γιατί ε, τα άρθρα στις εφημερίδες ε, αναφέρεται ότι ένας συνεργάτης φέρεται να είπε ότι ασκήθηκαν πιέσεις ώστε οι κανόνες ε, του, κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να παρακαμφθούν. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι συνέβη κάτι τέτοιο, ότι είναι ένα τέτοιο ενδεχόμενο, αλλά και αυτό πρέπει να το ψάξουμε. Οφείλουμε, γιατί αν κανείς ε, ε, διαμορφώνει τους κανόνες όπως θέλει, αλλήμωνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, έχω και άλλες ερωτήσεις, αλλά σταματώ προς το παρόν και ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ο συνάδελφος Μπορν είναι ο επόμενος. Ευχαριστώ, ε, κύριος Φων. Ε, ε, δεν θα ήθελα να μπω στο θέμα αυτό του προηγούμενου Προέδρου. Θα ήθελα να πω ορισμένα πράγματα πριν μπω σε κάποια άλλα ζητήματα. όσον αφορά τις κατηγορίες κατά του πρώην Προέδρου, θα ήθελα να πω σε σχέση με την απαλλαγή του 2014 την οποία αφορούν οι περισσότερες κατηγορίες. Τότε θα έπρεπε να το είχαμε κάνει όμως και όχι τώρα. Ε, ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποια ζητήματα που έχουν τεθεί και υπήρχαν και κάποια θέματα που έχουν ε, απευθυνθεί στο Γενικό Γραμματέα. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε πολύ σύντομα να λάβουμε τις σχετικές απαντήσεις. Ελπίζω ότι οι απαντήσεις αυτές θα μας δώσουν κάποιες διευκρινήσεις και κάποια, ε, κάποιες εξηγήσεις και θα μας καθησυχάσουν κάποιους για τα ζητήματα μηνύματα αυτά, γιατί δεν θα ανέμενα ε, ότι η διοίκηση του Κοινοβουλίου θα επέτρεπε κάτι το οποίο δεν ήταν σωστό και αν έχει γίνει κάτι τέτοιο στο παρελθόν, αυτό θέτει ζητήματα και για την ίδια τη διοίκηση. Ελπίζουμε λοιπόν μέχρι το τέλο αυτή τη εβδομάδα, αρχέ επόμενη, να λάβουμε τι απαντήσει για να μπορέσουμε κι εμεί να ε, τοποθετηθούμε. Και μετά μπορούμε τότε να μπούμε σε μια σωστή διαδικασία απαλλαγή. Ε, δεν νομίζω ότι θα μα κάνει κανένα καλό ούτε στην Επιτροπή του στο Κοινοβούλιο όταν συνδέουμε αυτό το πράγμα με άλλα ζητήματα ε, τα οποία είναι πολύ επίγοντα και για τα οποία πρέπει, στα οποία πρέπει να επικεντρωθούμε. Ε, δεν θέλω δηλαδή να συζητάμε γι' αυτό πριν από τι απαντήσει, ενώ εκκρεμούν άλλα ζητήματα πολύ σημαντικά. Ε, όσον αφορά την ευρύτερη εικόνα και την παρακολούθηση του, του προπολογισμού του Κοινοβουλίου, Υπήρχε ένα τμήμα εμπειρογνωμοσύνης που πρότεινε η ομάδα των Σοσιαλδημοκρατών να υπάρξει ε, για να δούμε ε, πώς είναι τα πράγματα ε, σε σχέση με τον προπολογισμό του Κοινοβουλίου. Δεν ξέρω αν αυτό είναι καλή ιδέα. Βλέπουμε πόσες περικοπές υπάρχουν. Καλό θα ήταν να δούμε μήπως υπάρχουν υφιστάμενες δομές που μας δίνουν τη δυνατότητα να το κάνουμε. Όσον αφορά τη διαφάνεια, όταν μιλάμε για διαφάνεια, συνήθως μιλάμε για τη διαφάνεια των γενικών, των, των εξόδων κίνησης ε, των γενικών επιδομάτων ε, και ε, από την άλλη πρέπει να εξασφαλίζουμε ότι δεν είναι τεράστιο το γραφειοκρατικό άχθος και ότι αυτό δεν δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στο σύστημα. Το σύστημα που χρησιμοποιείται από το Ηνωμένο Βασίλειο και την αντιπροσωπεία των ΛΥΜΠΕ ε, εμείς έχουμε έναν εξάρτητο ελεγκτή, ο οποίος έρχεται, δεν παίρνει πάρα πολύ χρόνο, ένα πρωινό να έρθει και να ρίξει μία ματιά το, στον τρόπο με τον οποίο αυτό το ε, επίδομα έχει χρησιμοποιηθεί. Ε, και τότε μπορεί να ε, πούμε ε, με βάση αυτήν την αξιολόγηση κατά πόσο έχει γίνει η σωστή χρήση ε, των ποσών αυτών και τότε να το, να το ανεβάζουμε στον ιστότοπό μας για να ξέρουν όλοι ότι τα χρήματα αυτά έχουν δαπανηθεί σωστά και ότι αυτό είναι αντικείμενο συμπεράσματος μιας, ενός ανεξάρτητου ελεγκτή. Δεν είναι τεράστιο έτσι το γραφειοκρατικό άχθος και ούτε το κόστος. Υπάρχουν τρόποι λοιπόν να είμαστε πιο διαφανείς. Μπορούμε να το κάνουμε με τέτοιο τρόπο που δεν δεν ε, προσθέτει στη γραφειοκρατία ούτε στο κόστος ε, του συστήματος. Ίσως θα μπορούσαμε να το δούμε και αυτό μια, ως μια πρόταση για να προχωρήσουμε. Ε, γιατί όλη την ώρα το συζητούμε. Κάτι ακόμη που θα ήθελα να θέσω όσον αφορά την έκθεση του κυρίου Ντε είναι το θέμα των γραφείων ενημέρωσης σε όλα τα κράτη-μέλη και κατά πόσο υπάρχει ανάγκη ύπαρξής τους. Κοιτάξτε, επειδή σκέφτομαι την ε, κατάσταση, την εκστρατεία με τον Brexit στο Ηνωμένο Βασίλειο, αν ο κόσμος δεν ήξερε απολύτως τίποτε, δεν ήξερε τίποτε για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, σίγουρα δεν ήξερε και πώς δουλεύει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, υπήρχαν γραφεία μόνο στο Λονδίνο και στη Σκωτία. Υπήρχαν τεράστια λοιπόν τμήματα του Ηνωμένου Βασιλείου, στα οποία δεν υπήρχε γραφείο πληροφόρηση. Οπότε εγώ δεν ξέρω κατά πόσο θα καλή ιδέα να μειώσουμε ε, ή να περιορίσουμε τα γραφεία αυτά. Για τα APAs τώρα, συμφωνώ με τον Τένις ότι χρειάζονται περισσότεροι ε, προστασία ειδικότερα ως προς τις καταγγελίες και ε, τις συμβάσεις που έχουν ε, τελικά ε, διακοπεί, να δούμε τι χρήματα λαμβάνουν όταν πηγαίνουν στο Στρασβούργο. Μπορεί να είναι πολύ χαμηλό το ποσό και είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθεί στέγαση με αυτά τα ποσά, για παράδειγμα. Πρέπει να, μπορούμε, να μπορούν να εξασφαλίζουν ότι είναι αρκετό το ποσό για να τους εξασφαλίσει και την ασφάλειά τους. Ξέρω ότι ο Γενικός Γραμματέας είπε ότι αυτό το θέμα θέμα εξετάζεται, όμως όσο περνάει ο καιρός, ε, τόσο ε, όσο και περισσότερο ε, πηγαίνουν οι άνθρωποι αυτοί στο Στρασβούργο, πρέπει να εξασφαλίσουμε το στομότερο δυνατόν θα λυθεί αυτό το ζήτημα κατά τις επισκέψεις στο Στρασβούργο. Ευχαριστώ. Συνάδελφε Ζάρ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όντω πολλά ενδιαφέροντα πράγματα εμπεριέχονται στο σχέδιο έκθεσης του κυρίου Ντεγιόγκα. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε διάφορα σημεία. Πρώτον, όλα αυτά που έχουν να κάνουν με τα πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα. Προτού αναφερθώ πιο συγκεκριμένα στα ζητήματα αυτά, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω λίγο τους κανόνες, τον κανονισμό και συγκεκριμένα τι λένε οι συνθήκες όταν διαβάζουμε και ακούμε διάφορα πράγματα για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και ιδρύματα, έχουμε με την εντύπωση ότι δεν έχουμε να κάνουμε με αξιοσέβαστους οργανισμούς. Εγώ νόμιζα ότι σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα, ένα πολιτικό κόμμα, ο οργανισμός θα πρέπει να είναι αξιοσέβαστος. Αντίθετα, έχουμε την εντύπωση ότι έχουμε να κάνουμε διεθνή μαφία. Και βέβαια, εγώ τίθομαι κατά της προσέγγισης αυτής. Σα υπενθυμίσω λοιπόν τι λένε οι συνθήκε και τι λέει ο κανονισμό. Στα πλαίσια μια δημοκρατία υπάρχουν συγκεκριμένοι δείκτε. Τώρα, το ότι υπάρχουν πολλά και διαφορετικά μάλιστα πολιτικά κόμματα είναι ένα πολύ σημαντικό δείκτη για την ύπαρξη τη δημοκρατία. Ο χάρτη των θεμελιδών δικαιωμάτων τη Ευρωπαϊκή Ένωση, στο άρθρο 12 και έχω μπροστά μου το κείμενο. Ο Βίκτορ Ιγκό, όπω ξέρετε, ο μεγάλος Γάλλος τογοτέχνης έλεγε ότι συμφωνούσε με το ζήτημα αυτό ότι όλοι έχουν το δικαίωμα να συνεδριάζουν, να συνέρχονται σε επίπεδο πολιτικό, συνδικαλιστικό. Σε ευρωπαϊκό μάλιστα επίπεδο οι συναντήσεις αυτές έχουν ως στόχο να προωθήσουν περισσότερο τη φωνή του Ευρωπαίου πολίτη όχι μόνο για να περάσει το επικρατέστερο μήνυμα, αλλά για να ακουστούν και όλες οι διαφορετικές απόψεις των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο χάρτης πολιτών δικαιωμάτων λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο προήμιό του λέει ότι βασίζεται κυρίως στις συνταγματικές παραδόσεις των κρατών μελών. Εγώ μεγάλος ευρωβουλευτής και ενδεχομένω συμφωνήσουν εδώ πέρα και κάποιοι Γάλλοι συνάδελφοι, στο άρθρο 4 του Γαλλικού Συντάγματο λέγεται το ακόλουθο. Τα πολιτικά κόμματα ασκούν τη δραστηριότητά του ελεύθερα, σε καθεστώ ελευθερία και ανεξαρτησία. Ο στρατηγό Ντεγκόλ είναι αυτό ο οποίο ε, συνέταξε το Σύνταγμα αυτό, μόνο ότι γνωρίζουμε ότι είχε μια συγκεκριμένη στάση, πολλέ φορέ συγκαταβατική απέναντι στα πολιτικά κόμματα, αλλά ήθελε και αυτός να θεσπίσει την απόλυτη ανεξαρτησία τους. Επίσης, η διάκριση των εξουσιών είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ σημαντικό. Δεν έχουμε Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, γι' αυτό το λόγο αντί να μιλάμε για διάκριση εξουσιών θα πρέπει να μιλάμε για ισορροπία εξουσιών στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν νομίζω όμως ότι χωρίς τις αρχές αυτές μπορούμε να μιλάμε πραγματικά για δημοκρατία και πολλές φορές μπορεί να υπάρχει μια περίεργη αιμομικτική θα λέγα, σχέση ανάμεσα σε οργανισμούς όπως η Όλαφ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο ίδιο πνεύμα, ανάμεσα στους δημοκρατικούς αν θέλετε δείκτες, τους πιο ουσιαστικού, το άρθρο 2 του εσωτερικού μας κανονισμού αναφέρεται το ότι ε, κάθε πίεση η οποία μπορεί να ασκηθεί στα πλαίσια μιας ε, εντολής ε, κοινοβουλευτικής δεν θα πρέπει να υφίσταται. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη. Ένα πολιτικό κόμμα, ένα σύλλογος, μία ομάδα πίεσης ή ακόμα και μία διοίκηση, ακόμα και αυτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν μπορεί να ασκεί πίεση σε έναν αυροβουλευτή κατά τη διάρκεια της εντολής του όσον αφορά την πολιτική τοποθέτησή του για παράδειγμα, όσον αφορά τις ε, υποχρεώσεις του, τι χρηματοοικονομικές σε σχέση με ένα πολιτικό κόμμα και όσον αφορά και την ίδια την οργάνωση της καθημερινής του εργασίας. Νομίζω θα έχουμε την ευκαιρία να επανέλθουμε στο ζήτημα αυτό. Όσον αφορά λοιπόν τα πολιτικά κόμματα θέλω να την θυμίσω απλώς κάποια πράγματα. Επίσης, στη διατύπωση που έχει επιλέξει ο συνάδελφος De Jong, και παραθετικά να πω ότι προφανώς γνωρίζω ότι έχει πάρα πολύ καλή εμπειρία, υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία με εκπλήσουν. Περνάω για παράδειγμα στα συμπεράσματά του, όπου θέτει το εξή ερώτημα. Αξίζει πραγματικά τον κόπο να συνεχίσουμε να χρηματοδοτούμε τα πολιτικά ευρωπαϊκά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα. Νομίζω ότι απάντησα στην ερώτηση αυτή μετά όσα είπα. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο προκαλεί εντύπωση. Όταν μας λέει ο κύριος Ντεγιόνκ ότι υπάρχουν ορισμένα πολιτικά κόμματα και ιδρύματα τα οποία έχουν παραπέσει σε σοβαρές παρατυπίες. Μα δεν μπορούμε να τους βάζουμε όμως στο ίδιο τσουβάλι, έτσι δεν είναι. Ξέρω ότι υπάρχουν ορισμένα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα τα οποία εντάσσονται στο δικό μου το κίνημα. Εγώ είμαι μέλος της Επιτροπής μας και επίσης ε, επικεφαλής πολιτικού κινήματος και δεν νομίζω ότι θα μπορούσαμε την παρατυπία αυτή, η οποία θα μου αφορούσε και εμένα, για 60.000 ευρώ για παράδειγμα, να θεωρηθεί ως σοβαρή αξιόπινη πράξη. Ξέρετε ότι το εθνικό μέτωπο στο οποίο συμμετέχω εμφανίζεται στο κίνημα αυτό το οποίο τίθεται να αμφιβόλω από τον εισηγητή στην έκθεση του αυτή ουσιαστικά μας λέτε ότι μόνο και μόνο επιμείς, επειδή εμείς καταβάλουμε μια χρηματοοικονομική συμβολή, ουσιαστικά χρηματοδοτούμε ένα εθνικό πολιτικό κόμμα. Μα το αντίθετο ακριβώς συμβαίνει. Το εθνικό μέτωπο ως εθνικό κόμμα είναι αυτό το οποίο χρηματοδοτεί το αντίστοιχο ευρωπαϊκό πολιτικό κίνημα. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει αν μη τι άλλο να διορθώσουμε τη διατύπωση σε κάποια σημεία στην έκθεση αυτή, διότι δίνονται λανθασμένες εντυπώσεις. Ο κύριος, ε, ο κύριος Βέλο, γενικός γραμματέας μας, μάλιστα σε προηγούμενη συνεδρίασή μας, είχε πει επιγραμματικά βέβαια ότι ε, η όλη αυτή η συζήτηση ήδη βρίσκεται ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι εναπόκειται στο δικαστήριο να αποφασίσει τελεσίδικα επ' αυτού. Σε κάθε περίπτωση, σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να δεχθώ εμείς ότι έχουμε υποπέσει σοβαρή αξιόπινη πράξη, όπως ουσιαστικά υπονοεί ο εισηγητής. Ακούσαμε για παράδειγμα τον Μαλτέζο Υπουργό Οικονομικών, ο οποίο μα μίλησε πριν από λίγο στην συνεδρίαση αυτή και ο οποίο είπε ότι το γενικότερο σφάλμα στο κοινοτικό προπολογισμό είναι 3,8%. Αυτό μειώθηκε στο 1% από κάποιον άλλο που πήρε το λόγο. Όταν όμως μιλάμε για 146 δισεκατομμύρια ευρώ, ακόμα και το 1% του ποσού αυτού ουσιαστικά αντιστοιχεί σε περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό ναι, αυτό όντως είναι σοβαρή παρατυπία που συνιστά αξιόπινη πράξη. Μολονότι όπω υπόθηκε σήμερα το πρωί, δεν μπορούμε να μιλάμε για απάτη, ενδεχομένω να υπάρχουν παρατυπίε οι οποίε είναι απλέ ατασταλείς, χωρί να αποτελούν απάτη. Αυτά. Τώρα, όσον αφορά την περίπτωση Σούλτ είναι αστείο να ακούμε τον άνθρωπο ο οποίο είχε μιλήσει τόσο πολύ για τη διαφάνεια να, υποπέ... να υποπίπτει ο ίδιο σε τέτοια σφάλματα κάθε φορά που οι πολιτικοί του αντίπαλοι ουσιαστικά προχωρούσαν σαν άλλες δραστηριότητε, πάντα δέχονταν τα πειρά του κυρίου Σούλτσα και αυτό δεν έχει να κάνει με τον προπολογισμό του 2009 και του 2010 Όσον αφορά το συγκεκριμένο πρόσωπο, πραγματικά νομίζω ότι ε, εδώ θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε και βέβαια η κατάσταση γίνεται αρκετά επονίδιστη για πάρα πολλούς που τον είχαν υποστηρίξει. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Θα πρέπει λοιπόν να θίξουμε το ζήτημα αυτό. Όσον αφορά τώρα το έργο και τη φύση της εργασίας των Ευρωβουλευτών, Ορισμένοι δίνουν την εντύπωση ότι ε, ο Ευρωβουλευτής ασχολείται μόνο με το νομοθετικό έργο. Το προπαρασκευαστικό έργο δεν είναι η μόνη αρμοδιότητα ενό Ευρωβουλευτή. Ένα Ευρωβουλευτή πρέπει να είναι σε επαφή με τα μέσα ενημέρωση, θα πρέπει να είναι σε επαφή επίση με τα εθνικά πολιτικά κόμματα πολλέ φορέ, γιατί καταλαβαίνετε ότι οι περισσότεροι συνάδελφοι έχουν ε, εκλεγεί με σύστημα αναλογικό. Ακόμα και ένας πρωτοετής φοιτητή γνωρίζει ότι το Εθνικό Πολιτικό Κόμμα είναι αυτό το οποίο μπορεί να καθορίσει τον, την εκλογή ενός ευρωβουλευτή ή όχι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι σαφώς το νομοθετικό έργο αποτελεί μία πτυχή της εργασίας μας, αλλά υπάρχει και όλη αυτή η έξω κοινοβουλευτική εργασία την οποία καλούμεθα να κάνουμε, όντας σε επαφή με τα εθνικά πολιτικά μας κόμματα και με τα μέσα ενημέρωσης όπως σας είπα. Σαφώς επίσης θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος για το έργο που κάνουμε όλοι μας, για το έργο που κάνουν οι διάφοροι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να διασφαλίσουμε τη σωστή χρησιμοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων, αλλά ας μην υπεργενικεύουμε, δεν θα πρέπει αυτή τη στιγμή προσπαθώντας να περισσώσουμε την κατάσταση ή να επιβάλλουμε διαφάνεια, να βάζουμε τα πάντα στην μια κοινή κατηγορία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να απαντήσω σε αυτό που είπε ο προηγούμενος ομιλητής για τα διαθέσιμα κονδύλια στα μέλη του Κοινοβουλίου και πώς δαπανώνται για να προσληφθούν διαπιστευμένοι βοηθοί. Ποια είναι τα καθήκοντά τους και τι μπορούν και τι δεν μπορούν να κάνουν οι βοηθοί και αν μπορούν να κάνουν δουλειά που θα έπρεπε κανονικά να γίνεται στο κράτος μέλος από το πολιτικό κόμμα. Αυτό βέβαια δεν εντάσσεται στη φετινή απαλλαγή, αλλά στο μέλλον πρέπει να το δούμε. Ο Σκιώδης μας μίλησε για, τις, για τη θέση της ομάδας και Ντένις, αν θέλεις να είναι πιο ε, αυστηρές οι προτάσεις για τα πολιτικά κόμματα και τα ιδρύματα, μπορούμε να δούμε τι πλειοψηφία θα υπάρξει. Τώρα, πολύ γρήγορα, για την παράγραφο 46. Τα γραφεία δηλαδή ενημέρωσης. Με σοκάρισε λίγο η παράγραφος αυτή, γιατί λες ότι κάποια γραφεία ενημέρωσης ίσως θα έπρεπε να κλείσουν και μιλάς συγκεκριμένα για Βρυξέλλες και Στρασβούργο. Εγώ είμαι Βέλγος, Φλαμανδός και αναφέρεσαι στο γραφείο ενημέρωση για το Βέλγιο, για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έτσι όπως είναι διατυπωμένη αυτή η παράγραφος, λέει ότι η ενημέρωση στο κοινό μπορεί να γίνει από το διαδίκτυο και όχι από γραφεία ενημέρωσης και να είναι και πιο αποτελεσματική ενημέρωση. Εμένα με ενοχλεί λίγο αυτό το πράγμα και με ανησυχεί γιατί δεν πιστεύω την αλήθεια. Αν δω τι κάνει το γραφείο ενημέρωσης του Βελγίου και ξέρω καλά, σας διαβεβαιώ ότι κάνουν πολλά περισσότερα, κάνουν πάρα πολλές δραστηριότητες και εκτός Βρυξελών φέρνουν γαλλόφωνους και ε, ε, φλαμαντόφωνους Βέλγους μαζί, ειδικού στην Ευρωπαϊκή ε, Ένωση, επιστήμονες και 22 Βέλγοι ευρωβουλευτές ε, αξιοποιούν όλους αυτούς τους ανθρώπους στις δραστηριότητες τους. Φαίνονται αυτά στους απολογισμούς και επίσης φαίνεται ότι ε, το μήνυμά τους και η ενημέρωση φτάνει σε πολύ ευρύτερα στρώματα από ό,τι μπορούμε να κάνουμε από το Κοινοβούλιο. Υπάρχει προστιθέμενη αξία λοιπόν στο Γραφείο Ενημέρωσης του Βελγίου, το οποίο βρίσκεται εδώ πολύ κοντά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπάρχει πραγματικά προστιθέμενη αξία και το βλέπω στην πράξη και δεν νομίζω ότι μπορεί να αντικατασταθεί από καλύτερη πρόσβαση στο διαδίκτυο και περισσότερες δυνατότητες γιατί είναι άλλου τύπου δουλειά αυτή. Οπότε εδώ οπωσδήποτε εγώ θα καταθέσω σχετική τροπολογία για να αναδιατυπωθεί τουλάχιστον η παράγραφος αυτή. Συμφωνώ ότι αν δούμε ε, ευρύτερα τα γραφεία ενημέρωσης και λάβουμε υπόψη μας ε, ότι συχνά ο κόσμος ε, αντιμετωπίζει επικριτικά το Κοινοβούλιο και τα άλλα θεσμικά όργανα, σίγουρα θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας αυτό όταν κρίνουμε τα γραφεία ενημέρωσης. Αλλά τα γραφεία ενημέρωσης δεν πρέπει να είναι το τμήμα προπαγάνδας πρέπει να κάνουν ενημέρωση. Αυτό είναι το καθήκον τους. Να διαβεβαιώνουν ότι ενημερώνουν το κόσμο για το πραγματικό έργο που γίνεται στα θεσμικά όργανα και στο κοινοβούλιο προκειμένου. Δεν ξέρω τι κάνει το γραφείο ενημέρωση στο Στρασβούργο, αλλά ξέρω πολλά για το βελγικό γραφείο. Και δεν θα το κλείνα. Δεν θα το παραμέριζα δηλαδή με σε μία παράγραφο στην έκθεση De Jong. Όσοι με ξέρουν, ξέρουν ότι κάθε άλλο παρά Βέλγος εθνικιστής είμαι. Είμαι πολύ ευρωπαϊστής, φιλοευρωπαίος, παρόλο που βλέπω κριτικά την Ευρώπη. Πάντως το, και το Βελγικό Γραφείο Ενημέρωσης πολλές φορές ε, ενημερώνεται και από μένα. Και εάν ε, δω ότι προπαγανδίζει πράγματα, αυτό το στιγματίζω. Η συνάδελφος Αγιάλα Ζέντερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε. Όσον αφορά τον πρώην πρόεδρο του ε, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εγώ καθυστέρησα να έρθω αλλά υπάρχουν συνεργάτες του ε, εστιατορίου που τους γνωρίζουμε εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα και μας ζήτησαν να είμαστε εκεί για να τους αποχαιρετήσουμε επειδή έφευγαν. Συμφωνώ με τη γενική ουσία όσον αναφέρει ο κύριος De Jong στην ε, έκθεσή του. Παρακολούθησα και την επιχειρηματολογία του κυρίου Γκάγερ σε σχέση με το ζήτημα του πρώην Προέδρου με τα νέα τα οποία προέκυψαν ε, τον Απρίλιο πριν από τις εκλογές και επανέρχονται τώρα. Δεδομένου ότι τώρα τα πράγματα παίρνουν τις διαστάσεις ε, αυτές, εμείς διερωτώμεθα μήπως ε, ο ελεγκτής των ε, δεδομένων θα πρέπει να συνεργαστεί μαζί μας για το θέμα αυτό. Ε, ο εισηγητής υποβάλλει μια σειρά προτάσεων. Δεν αμφιβάλλω για τις καλές τους προθέσεις όσον αφορά το στόχο της διαφάνειας, αλλά πρέπει κάποια δεδομένη χρονική στιγμή να αναρωτηθούμε πώς η απόλυτη διαφάνεια συνάδει με την προστασία του ιδιωτικού βίου και των προσωπικών δεδομένων. Ε, πρέπει να ε, είμαστε υπόλογοι και κάθε μέρα, αλλά και κάθε πέντε χρόνια στους ψηφοφόρους μας, αλλά και ε, στο προσωπικό με το οποίο συνεργαζόμαστε. Το προσωπικό μας όμως δεν πρέπει υποχρεωτικά να ακολουθεί τη δική μας μοίρα. Υπάρχουν κάποια προβλήματα τα οποία μπορεί να έχουμε εμείς ε, με το προσωπικό μας και ε, θα έπρεπε βέβαια να γίνουν προτάσεις σε σχέση με τους βοηθούς μας. Εγώ θα υποβάλω και σχετικές τροπολογίες Νομίζω ότι πρέπει να αποσαφηνίσουμε το πλαίσιο της προστασίας των δεδομένων όσον αφορά το περιβάλλον μας. Και δεν μιλάω μόνο για τους ε, ευρωβουλευτές, μιλάω για τους βοηθούς κλπ. Για το βραβείο Λουξ τώρα. Κάποιες ε, κριτικές ε, είχαν ε, ακουστεί. Ε, εγώ βλέπω τις ταινίε και ψηφίζω. Είχαμε δει ότι οι ταινίε που παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο του βραβείου Λουξ φέτος ε, είχαν επιτυχία και σε σημαντικά φεστιβάλ κινηματογράφου. Πρέπει λοιπόν να υπερασπιστούμε ταινίε οι οποίες έχουν σχέση με τις ευρωπαϊκές αξίες. Όταν βλέπουμε ότι αυτό επιτρέπει σε κάποιες ταινίε να περάσουν από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού και να φτάσει στη μέκα του κινηματογράφου ε, σήμερα, ε, μου φαίνεται λογικό ως επιχείρημα για να υποστηρίξουμε τους συγκεκριμένους ε, σκηνοθέτες. Είναι κάτι το οποίο ε, υπερβαίνει βέβαια την νομοθετική δημοσιονομική μας ε, δραστηριότητα. Όσον αφορά τώρα τη διαχείριση του Κοινοβουλίου, νομίζω ότι πρέπει να επιστήσουμε την προσοχή μας ε, σε ε, σχέδια που ε, έχουν δρομολογηθεί εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, ε, πράγματα που εδώ και καιρό τα συζητούμε, τα κτίρια, το PRS λόγω της ελαστικότητας του προϋπολογισμού μας, το θέμα της ποιότητας της εργασίας μας. Πιστεύω εν ότι θα μπορούσαμε να ξανακάνουμε μία ενημέρωση, έναν απολογισμό των μεγάλων ε, προγραμμάτων που τα είχαμε αφήσει κάπως σε και τα οποία θα έπρεπε ενδεχομένως ε, να ξαναπάρουν μπρο και να επιταχύνουν κάπως. Όσον αφορά τώρα την απαλλαγή για το 2015... Λοιπόν, και εγώ να πω. Μακάρι να ίσχυε αυτό που είπε ο κύριος Ντεγιόγκ ότι ό,τι το είπαμε δεν το ξαναλέμε. Γιατί δεν θα, λέγαμε και θα ξαναλέγαμε τις, για τις έδρες. Αλλά πολλές φορές ε, χρειάζεται αυτό στην απαλλαγή. Τώρα αν δούμε τον πρώην πρόεδρο, αυτά που έχουμε τώρα είναι καινούργια στοιχεία. Το 2014 δεν τα είχαμε ούτε στις παραγράφους που αφαιρέθηκαν τότε κατά την ψηφοφορία. Δεν υπήρχαν όλα αυτά και επειδή είναι καινούργια στοιχεία και επειδή ε, τεκμηριώνονται και ακόμα δεν, τα έχουμε δει όλα, οπωσδήποτε θα πρέπει να αναφερθούν αντικειμενικά προφανώς. Σύμφωνα απόλυτα με τον συνάδελφο Γκάιερ και με τον συνάδελφο Ντε Εδώ πρόκειται για την αξιοπιστία και πρέπει να πω ότι ανεξάρτητα από το πολιτικό χρώμα του Προέδρου θα έπρεπε να εξετάσουμε τα θέματα αυτά του τύπου. Το θέμα τώρα των ταξιδίων αυτών μεγάλης διάρκειας. Ενδιαφέρον το ερώτημα, το έχουμε ξαναθέσει το 2013, νομίζω το 12, το 2013, μας είχε πει η διοίκηση ότι στο μέλλον δεν θα γίνονται μακράς διάρκειας υπηρεσιακά ταξίδια γιατί είναι πολύ ακριβά. Τώρα το γερμανική, η γερμανική υπηρεσία τύπου λέει ότι είναι οικονομικά τα ταξίδια αυτά. Αντίφαση, συνάδελφε Σμιτ. Θέλω να μάθω λοιπόν τι ισχύει. Υπάρχουν 13 ε, υπάλληλοι που κάνουν αυτή τη στιγμή ε, είναι σε τέτοιο ταξίδι. Και οπωσδήποτε πρέπει να κάνουμε ερωτήσεις σχετικά. Εμείς έχουμε το σχετικό καθήκον οι κανόνες μας πολλές φορές ε, επιδέχονται μιας πιο ευρείας διερμηνίας. Θα πρέπει όμως να δούμε. Μπορεί κάποιος να πάει και να εγκατασταθεί εκεί στη... Ε, και τα Σαββατοκύριακα να, μην... να μένει εκεί και να μην επιστρέφει ποτέ. Ε, όλα αυτά θα πρέπει να τα δούμε ο επαγγελματική, η επαγγελματική έδρα είναι οι Βρυξέλλες. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν πώς υπολογίζονται σε αυτές τις περιπτώσεις ε, επιδόματα, αποζημιώσεις κλπ. Ε, υπάρχουν κριτήρια για να δούμε αν όντως χρειάζεται το υπηρεσιακό ταξίδι. Αν υπάρξουν ε, ανάγκες για να παρέμβουμε θα το κάνουμε όπως κάναμε και στο παρελθόν. Λοιπόν, θα το δούμε με κάθε αντικειμενικότητα το θέμα. Πρέπει και θα το κάνουμε, γιατί αυτό έχει να κάνει με την αξιοπιστία μας. Τώρα, για τα γραφεία ενημέρωση του Κοινοβουλίου, τα έθιξαν πολλοί συνάδελφοι και με κάποια έκπληξη ε, είδα ότι εξετάζουμε και την νομιμότητά τους. Ε, δεν είχαμε ασχοληθεί με αυτό το θέμα μέχρι τώρα. Αν έχουν προκύψει, γιατί δεν υπήρχαν στοιχεία. Αν υπάρχουν στοιχεία ε, θα πρέπει να τα δούμε. Δεν ξέρω αν είναι τόσα πολλά ώστε να δικαιολογούν ένα τόσο μεγάλο βήμα που θα ήταν η πρόταση για να κλείσουν ορισμένα. Ε, πρέπει να δούμε ποιες είναι οι αδυναμίες. Τώρα, για το κώδικα διοντολογίας των μελών και την ομάδα εργασίας, η ελευθερία της εντολής είναι σημαντική. Και εμείς ε, έχουμε διαφορετικά καθήκοντα ως πολιτικοί. Και βεβαίως ως βουλευτής ε, δεν θέλω να δώσω όπλα που θα χρησιμοποιηθούν εναντίον μου αν, ε, αν παρακαλέσουμε την ε, διοίκηση να ορίσει τι προβλέπει η κοινοβουλευτική εντολή, αλλήμωνό μας. Ε, αυτό over my dead body όπως λέμε. Ε, γιατί υπάρχει κίνδυνος να γίνει αυτό αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης. Βέβαια υπάρχει μεγάλη διαφορά, τεράστια διαφορά μεταξύ αυτού που συζητούμε ε, για τον πρώην πρόεδρο και το, φρον, ε, το εθνικό μέτωπο. Ε, χωρίς να θέλω να υπερασπιστώ τον πρόεδρο, νομίζω ότι οι κανόνες ε, σχετικά με το πώς θα γεννηθεί κάποιος συνεργάτης του Εθνικού Μετώπου, κάθε, κάθε κόμματος ή πολιτικής ομάδας είναι ξεκάθαρη και εδώ δεν υπάρχουν αμφιβολίες. Αυτά ήθελα να πω και καλό είναι τώρα να πάρει το λόγο Ντένις και να κλείσει το θέμα. Ευχαριστώ Ίγκε. Θα προσπαθήσω να συνοψίσω λίγο τις παρατηρήσεις μου ώστε να είμαι σύντομος. Αναφέρθηκαν ε, ορισμένα ζητήματα από αρκετούς συναδέλφους, το ζήτημα της διαφάνειας, καθώς επίσης και το ζήτημα που έχει να κάνει με την γενική αποζημίωση των ευρωβουλευτών. Έλαβα email πρόσφατα από διάφορους ψηφοφόρους οι οποίοι μου λέγανε ότι δεν πρόκειται να σας ξαναψηφίσουμε γιατί πέρα από το μισθό σας λαμβάνετε κάθε μήνα και 4.000 ευρώ επιπλέον. Και οι άνθρωποι αυτοί μου λέγανε ότι αν δούμε το επίπεδο φτώχεια στην ε, Ολλανδία, τα χρήματα αυτά θα μπορούσαν να πανηθούν, με συγχωρείτε με καλύτερο τρόπο. Εγώ του είπα ότι ένα πολύ μεγάλο μέρο των αποδοχών μου τα επιστρέφω ουσιαστικά στη χώρα μου. Πάντω, σε τακτική βάση, στις κάτω χώρες, βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά άρθρα στον τύπο για το ζήτημα του General Allowance, της γενικής αυτής αποζημίωσης των ε, Ευρωβουλευτών. Αν πραγματικά λοιπόν θέλουμε να ανταποκριθούμε σε αυτή την επίκριση η οποία πάρα πολλές φορές είναι δικαιολόγητη τελικά, αν μη τι άλλο πετείται ένας χι βαθμός διαφάνειας. Θα μπορούσαμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αυτό με διάφορους τρόπους και ενδεχομένως στο τέλος της θητείας των Ευρωβουλευτών θα μπορούσε να γίνεται και ένα συνολικός έλεγχος. Δεν λέω ότι θα πρέπει να κοινοποιούμε οποιαδήποτε απόδειξη αγοράς. Θα πρέπει πάντως να αποσαφηνίσουμε προς τους ε, Ευρωπαίους πολίτες ότι γίνονται έλεγχοι των δαπανών μας. Εγώ στην έκθεση αναφέρομαι στη διοίκηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ζήτημα ανοιχτό προς συζήτηση. Μία άλλη εναλλακτική θα ήταν ένα μέρος της γενικής αποζημίωσής σας να χρησιμοποιηθεί για να πληρωθεί ένας εξωτερικός ελεγκτής, ο οποίος θα κάνει αυτόν τον έλεγχο. Με τον ένα τον άλλο τρόπο θα πρέπει να αποσαφηνίσουμε προς Ευρωπαίους πολίτες ότι δεν πρόκειται για έναν επιπλέον μισθό. Είναι ένας χρηματοδοτικός φάκελος που έχουμε για να καλύπτουμε διάφορες δαπάνες. Δεν νομίζω λοιπόν ότι ε, πηγαίνω πάρα πολύ μακριά με τις ε, παρατήρησει που κάνω. Αυτό που λέω είναι ότι ο έλεγχος αυτός θα πρέπει να γίνεται με τρόπο αποτελεσματικό. Δίνω απλώ κάποια παραδείγματα για το πώς θα μπορούσε να γίνει αυτός ο έλεγχος, ενδεχομένω να αφορά δαπάνε από ένα κατόφλι και πάνω και προτείνω ποιο θα μπορούσε να κάνει, ένα εξωτερικό ελεγκτή για παράδειγμα, ποιο θα μπορούσε να κάνει τον έλεγχο αυτόν. Μα είχε απασχολήσει το ζήτημα αυτό και πέρυσι. Εγκρίναμε σχετική πρόταση στη σχετική έκθεση απαλλαγή στην Ολομέλεια. Είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάντω. Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα που έδειξαν πολλοί συνάδελφοι είναι η κατάσταση που έχει προκύψει με τον πρώην πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τι ενδεχόμενε παρατυπίε τι οποίε να έχει υποπέσει. Η σημερινή συζήτηση ήταν πάρα πολύ χρήσιμη, γιατί από ό,τι φαίνεται όλοι συμφωνούμε ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αντικειμενικά. Και ουσιαστικά όλοι θέλουμε η διοίκηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να απαντήσει στα ερωτήματά μας. Ελπίζω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε μια συζήτηση για το ζήτημα αυτό και με τους σκιώδεις συγητές. Το πρόβλημα είναι ότι ε, το Μάρτιο κατά τη διάρκεια τη εβδομάδα στο Στρασβούργο. Εμεί θα έχουμε εθνικέ εκλογέ στις κάτω που μόνο δεν θα καταφέρω να έρθω στο Στρασβούργο εκείνη την εβδομάδα ή τουλάχιστον θα έρθω για ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Πάντω, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να καταφέρουμε να δούμε πώ θα αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αυτό, εμπίπτει στι αρμοδιότητε τη δική μα επιτροπή και θα πρέπει να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα και σε συγκεκριμένε συστάσει οι οποίε θα εμπλουτίσουν περισσότερο αυτή την έκθεση. Τώρα, όσον αφορά τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα. Δεν κατάλαβα πολύ καλά αυτά που υπόθηκαν για μένα και για την έκθεσή μου. Σε καμία περίπτωση δεν αναφέρω ότι είμαι κατά των επιδοτήσεων. Στη συγκεκριμένη αυτή παράγραφο λέω απλώ ότι θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση για αυτό το 15% επιπλέον εσόδων δώρων, δωρεών μπορούμε να πούμε, που δέχονται ή που μπορούν να έχουν τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα. Ουσιαστικά αυτό που λέω είναι ότι θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε λίγο το σημείο αυτό. Το Προεδρείο του Κοινοβουλίου συζητά το ζήτημα αυτό και μάλιστα έχει προτείνει να μειωθεί το σχετικό κατόφλι χρηματοδότηση. Εγώ δεν είπα ότι θα πρέπει να καταργήσουμε τι επιδοτήσει στα κόμματα. Το αντίθετο. Αν το ποσοστό αυτό τελικά μειωθεί στο 5%, τότε οι επιδοτήσει μπορούν να ανέλθουν στο 95%, ενώ αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο 85% των δαπανών. Επομένω, σε καμία περίπτωση δεν είχα την πρόθεση να πω αυτά τα οποία είπε ο συνάδελφο. Για κάποια άλλα σημεία τώρα, όσον αφορά του βοηθού των Ευρωβουλευτών, και όσον αφορά τον τρόπο που προστατεύουμε τους καταγγέλτες, συμφωνώ με τους πράσινους στο σημείο αυτό. Προσπάθησα να καταλήξω σε ένα καλό κείμενο, αλλά προσβλέπω και στις δικές σας τις παρατηρήσεις για να βελτιωθεί το σχετικό κείμενο. Και ο κύριος Ντέρεκ Βόουν επίσης έκανε κάποιες παρατηρήσεις. Όσον αφορά τις δαπάνες για τους βοηθούς μας στο Στρασβούργο, οι δαπάνες αυτές διαφέρουν από τις δαπάνες του υπόλοιπου προσωπικού. Αν πραγματικά θέλουμε να καλύψουμε τους ανθρώπους αυτούς και για την ε, διαμονή τους στο Στρασβούργο, θα πρέπει το ποσό αυτό ε, να αυξηθεί. Το ποσό το οποίο δίνεται αυτή τη στιγμή είναι το ελάχιστο δυνατό προκειμένου να μπορεί κανείς να διαμείνει στο Στρασβούργο. Το Προεδρείο πάντως εξετάζει περαιτέρω το ζήτημα αυτό. Όσον αφορά τώρα τις, τα γραφεία ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεν νομίζω ότι θα πρέπει απλώ να φερθούμε εδώ πέρα στα γραφεία αυτά καθε αυτά και ουσιαστικά δεν ήθελα να πω εγώ κάτι τέτοιο στην εκθεσή μου και αναφερόμουν περισσότερο στα γραφεία ενημέρωση που έχουμε στι Βρυξέλλε και στο Στρασβούργο και όχι τόσο πολύ στα υπόλοιπα κράτη-μέλη τη ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο συνάδελφο που έθεσε το ζήτημα αυτό δυστυχώ χρειάστηκε να αποχωρήσει. Θα ήθελα να μιλήσω διμερό μαζί του για να αποσαφηνίσω το σημείο αυτό. Το πιο σημαντικό είναι να καταφέρουμε να έχουμε μεγαλύτερη άμεση επαφή με τον απλό Ευρωπαίο πολίτη. Νομίζω ότι αυτό δεν επιτυγχάνεται αυτή τη στιγμή από τα γραφεία ενημέρωση, τα οποία έρχονται σε επαφή με ευρωβουλευτέ, με φοιτητέ, με καθηγητέ που ήδη εξορισμού ενδιαφέρονται για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί επικεντρώνονται περισσότερε δραστηριότητέ του. Σαφώ χρειαζόμαστε και του ανθρώπου αυτού, αλλά χρειαζόμαστε και προγράμματα ενημέρωση, πολιτικέ επικοινωνίε, οι οποίε θα φτάνουν και σε ανθρώπου οι οποίοι είναι επικριτικοί για την Ευρωπαϊκή Ένωση. θα μπορούσαμε κατά αυτόν τον τρόπο να επιλύσουμε και όλες αυτές τις παράνοιες που υπάρχουν, παρανοήσεις με συγχωρείτε, σε σχέση με την αποζημίωση των ε, ευρωβουλευτών. Μέσω της άμεσης αυτής επαφής που θα μπορούσαμε να έχουμε με τους Ευρωπαίους πολίτες, μέσω των γραφείων ενημέρωσης, θα μπορούσαμε να διασκεδάσουμε τυχόν ανησυχίες που υφίστανται στους Ευρωπαίους πολίτες. Όσον αφορά αυτά που είπε ο συνάδελφο από του φελεύθερους για την κατάρτιση και την τεκμηρίωση και ότι θα πρέπει και εκεί να έχουμε προπολογισμό βάση επιδόσεων. Σαφώ θα πρέπει και εδώ πέρα να καταμετρήσουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Σε καμία πάντω περίπτωση δεν πρέπει να δημιουργήσουμε μία υπηρεσία η οποία θα πρέπει να παράγει πάρα πολύ σημαντικό έργο μόνο και μόνο για να το πουλήσει σε εμά και να πούμε εμεί ότι όντω ναι, κοιτάξτε, έχει πολύ καλέ επιδόσει. Προφανώ οι υπηρεσίε αυτέ θα πρέπει να τα αποκρίνονται στι πραγματικέ μα ανάγκε και αν συνταχθούν οι σχετικές εκθέσεις, τότε θα πρέπει να γίνεται και μια κάποια ανάλυση της εργασίας αυτών των υπηρεσιών, όπου να μπορούμε να θίξουμε συγκεκριμένα στοιχεία και να τα ποσοτικοποιήσουμε επίση ω προς τις δαπάνες. Χρειαζόμαστε πάντως την υπηρεσία αυτή για την υποστήριξη του δικού μας του έργου. Ε, 6 Μαρτίου, 2 η ώρα το μεσημέρι, προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών. Τελειώσαμε με το 58. Προχωρούμε στο 59, σημείο της ημερήσιας διάταξης, απαλλαγή 2015. Ο συνάδελφος ο Μαρζέ θα λάβει μέσα στο λόγο ως εισηγητής. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Παρακαλώ όσοι θέλουν να αποχωρήσουν, να αποχωρήσουν σύντομα. Euh, θα παρουσιάσω τώρα την έκθεση σε σχέση με την ε, απαλλαγή για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. Θα ήθελα να πω ότι αυτό το σχέδιο έκθεσης ήταν αντικείμενο μακράς εργασίας, ε, μακροχρόνιας, ε, λεπτομερούς, ε, εμπεριστατωμένης. Είχα πολλές ε, συνεδριάσεις εργασίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που την ευχαριστώ για τη διαθεσιμότητά της ειδικότερα τον Επίτροπο Μίτσα τον οποίο ε, γνώρισα και θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω το σύνολο των ε, συναδέλφων τους οποίους συμπεριέλαβα από τη στιγμή της σύνταξης του κειμένου, τους κοιόδης εισηγητές, αλλά και τους συντάκτες γνωμοδότησης των άλλων ε, επιτροπών που γνωμοδότησαν. Έχετε στη διάθεσή σας ε, την πρόταση κειμένου. Δεν θα μπω συνεπώς σε λεπτομέρειες για όλες τις προτάσεις που διατυπώνω. Θα ήθελα όμως ε, να ε, τονίσω αρκετά κεντρικά σημεία τα οποία αναδύονται από την έκθεσή μου και έχουν άμεση σχέση με το δημοσιονομικό έλεγχο. Θα ήθελα λοιπόν καταρχάς να αναφερθώ στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αξιοπιστία των ε, ταμείων και τη δήλωξη αξιοπιστίας της ΔΕΒΚΟ. Για το 2015 υπενθυμίζω ότι αφορούν ε, το 8ο, 9ο, 10ο και 11ο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης ε, και υπήρξαν τέσσερις μέθοδοι εφαρμογής. Στην έκθεση βλέπετε ότι επικροτώ τις προσπάθειες που κατέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη μείωση ε, των προηγούμενων προχρηματοδοτήσεων, ε, των ε, υπολείπων προς καθάριση και των συμβάσεων που εξέπνεαν. Όμως, θεωρώ θλιβερό έλλειψη, την έλλειψη πληρωμών του 2015 που οδήγησαν σε προβλήματα δημοσιονομικά όσον αφορά την κανονικότητα των λογαριασμών. Δυστυχώς δεν έχει πέσει το ποσοστό σφάλματο ε, από το 2014, 3,8%. Αντιθέτως αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια. 25% των πληρωμών που ανέλησε το ελεγκτικό συνέδριο ε, βρέθηκαν ότι είχαν σφάλματα και ότι η τυπολογία των σφαλμάτων παραμένει ίδια. Θα ήθελα λοιπόν να επιστήσω την προσοχή της Επιτροπής ακόμη περισσότερο για τέτοιου είδους σφάλματα, ειδικότερα για το μέλλον ε, και απουσία των δικαιωμάτων δικαιολογητικών, όπως επίσης και μη σεβασμό των ε, κανόνων της ιστορικής αγοράς όσον αφορά την ανάκτηση, την ανάκτηση των ε, φόρων ε, προχρηματοδότησης. 9,6 εκατομμύρια ευρώ προχρηματοδότησης που δεν χρησιμοποιήθηκαν ε, εσφαλμένως ενεγράφησαν ως επιχειρησιακά προϊόντα και νομίζω ότι η Επιτροπή πρέπει να λάβει νέα μέτρα ώστε να μην υπάρξουν τέτοιου είδου σφάλματα στο μέλλον, γιατί ουσιαστικά πρόκειται για την ακαιρεότητα των ενωσιακών κονδυλίων, ε, αλλά ε, δεν ε, μπορώ να παραγνωρίσω και την πρόοδο που σημειώθηκε όσον αφορά την, τους φόρους ε, προχρηματοδότησης. Θα μπορούσαμε να μπούμε και σε περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά τους ε, εκτονιστέρων των ε, ελέγχους και εδώ υπάρχουν κενά ελέγχων και ζητώ από την Επιτροπή να διορθώσει αυτά τα σφάλματα. Να υπογραμμίσω επίσης ότι σύμφωνα με το ελεγκτικό συνέδριο η Επιτροπή θα μπορούσε να είχε μειώσει το ποσοστό σφάλματος κατά 1,7% αν είχε χρησιμοποιήσει όλες τις πληροφορίες που είχε στη διάθεσή της. Όσον αφορά τώρα τα στοιχεία που έχουν να κάνουν με το πλαίσιο της αξιοπιστίας, εδώ χαίρομαι ε, που η Επιτροπή ακολούθησε τις συστάσεις ε, του Κοινοβουλίου ε, με διάφορα αποθεματικά διαφορετικά και όχι ένα γενικό αποθεματικό. Υπενθυμίζω και ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει υπόψη τις δράσεις που έχουν δρομολογηθεί για το κάθε αποθεματικό. Όσον αφορά το African Peace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 Ε, κάναμε μία συζήτηση και κλεισμένων των θυρών και ευχαριστώ την Πρόεδρο όπως επίσης και την Πρόεδρο της Επιτροπής Ανάπτυξης που διοργάνωσαν αυτή τη συζήτηση που ήταν πολύ ενδιαφέρουσα που μας έδωσε τη δυνατότητα να θέσουμε ερωτήματα να τονίσουμε τις ε, δικές μας ανησυχίες και να λάβουμε μία σειρά απαντήσεων από πλευράς ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής απαντήσεων που κατά την άποψή μου ακόμη παραμένουν ανεπαρκείς. Αναμένω ε, επομένως ε, και υποθέτω ότι και οι συνάδελφοι θα συμφωνήσουν μαζί μου ε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δράσει συγκεκριμένα προκειμένου να προσαρμοστεί η διακυβέρνηση και οι ευθύνες οι αντίστοιχες των εμπλεκομένων φορέων για την παρακολούθηση του μέσου αυτού και κυρίως ε, να ε, ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις διορθωτικές ε, ενέργειες που θα γίνουν και που πρέπει να γίνουν όπως επίσης και για την ανάκτηση των ποσών και τις μελλοντικές βελτιώσεις. Δεύτερο σημαντικό σημείο σε σχέση με την έκθεσή μου. Ε, θέλησα, θα το είδατε, να υπερισχύσει μια προσέγγιση προσανατολισμένη προς τα αποτελέσματα και ε, την αναζήτηση των επιδόσεων και διατυπώνω κάποιες προτάσεις ε, για τη βελτίωση των επιδόσεων και της αποτελεσματικότητας για τη διαχείριση του ΕΤΑ. Υπάρχουν πάρα πολλές προτάσεις, δεν πρόκειται να τις απαριθμίσω λεπτομερώς, θα ήθελα απλώς να επιμείνω στην πρόταση ανάπτυξης μιας τυπολογίας ε, αιτιών ε, μπλοκαρίσματος και των ε, δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι αντιπροσωπείες για την εφαρμογή των προγραμμάτων, όπως επίσης και υποχρέωση άμεσης ενημέρωσης αυτή τη στιγμή ε, έχει ταξινομηθεί ως κόκκινο τρεις φορές, τρεις ε, συνεχόμενες χρονιές ένα πρόγραμμα και να προβλέψουμε ε, ως τελευταία λύση την αναστολή των πληρωμών με βέβαια απόφαση του δικαστηρίου και τελευταία πρόταση ε, που είναι αυτονόητη και αφορά το σύνολο των ευρωπαϊκών πολιτικών και βεβαίως και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης ε, είναι η απαραίτητη απλοποίηση των κανόνων ελέγχου απαραίτητον για να μειωθεί το ποσοστό σφάλματος. Τρίτο, τρίτη μεγάλη πτυχή αφορά τους ε, εξωτερικούς ε, ε, φορείς, οι οποίοι όμως συμμετέχουν στους στόχους της πολιτικής αυτής. Τα καταπιστεύματα, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τις, ε, τους διεθνείς οργανισμούς. Θα διαβάσατε την έκθεση, ε, διαπιστώνεται ότι αυτό δημιουργεί ε, σειρά προβλημάτων ως προς τον έλεγχο και για τα trust funds, τα καταπιστεύματα και για την ΕΤΕΠ και ε, για τους διεθνείς οργανισμούς. Ε, νομίζω ότι μπορούμε παράλληλα να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε δύο στόχους, μεγαλύτερη διαφάνεια, ε, καλύτερος έλεγχος και παράλληλα έλεγχος των πολιτικών στόχων εφόσον κάθε εξουσιοδότηση συμμετέχει στους πολιτικούς στόχους που έχουμε ορίσει. Τέλος, θα ήθελα να επιμείνω επί κάποιων ε, γενικών ε, σημείων που είναι κάπως πιο πολιτικά ε, και αφορούν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. Είμαστε εδώ στην Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμών και μας ανησυχεί πάρα πολύ το ζήτημα των επιδόσεων. πολύ ε, θεμητά νομίζω, ε, διερωτώμεθα, ε, έχουμε κάποια ερωτηματικά για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας, αναπτυσσικής βοήθειας. Έχουμε κάποια ερωτηματικά σε σχέση με την συνοχή του συνόλου των ευρωπαϊκών πολιτικών, γιατί βλέπουμε δυστυχώς ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι προσπάθειες που καταμβάλλονται από τους υπεύθυνους της πολιτικής αυτής ε, αποδυναμώνονται, υπονομεύονται από την εφαρμογή άλλων πολιτικών και αναφέρομαι στην εμπορική πολιτική, αναφέρομαι στην αλλιευτική πολιτική επί αλλά θα μπορούσαμε να αναφέρουμε και πολλούς άλλους ε, τομείς υπάρχει μια πραγματική ανάγκη να υπάρξει μια συνοχή και να ε, σκεφτόμαστε λίγο πιο σφαιρικά. Επίσης θα ήθελα να επιμείνω ε, στο γεγονός και όλοι το, είπατε, ε, το είπαν αυτό και στην συζήτηση την προηγούμενη φορά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η αναπτυξιακή πολιτική επηρεάζεται ε, και από ε, κάποιες κρίσεις ε, οι οποίες μπορεί να ακυρώσουν ή να μετριάσουν την επίτευξη των στόχων. Εγώ είμαι από μία άκρος απομακρυσμένη περιοχή ε, και ξέρω ότι στη Σακέ για παράδειγμα αν υπάρχει μια θεοπινία, ένας κυκλώνας ε, ε, εξαιρετικής έντασης, προσπάθειες ετών ακυρώνονται. Το ίδιο ισχύει και όταν υπάρχει μια πολιτική κρίση ή ένας πόλεμος. Πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη κατά την αξιολόγηση που κάνουμε της ε, πολιτικής αυτής της αναπτυξιακής. Τρίτο σημείο το οποίο με απασχολεί όλος ιδιαίτερος και είχα την ευκαιρία να το συζητήσω με τον Επίτροπο Μίτσα ε, στην Αρούμπα ε, πριν από 10 μέρες για το Φόρουμ Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, υπερποντίων χωρών και εδαφών είναι το θέμα ε, των υπερποντίων χωρών και εδαφών έχουν ε, συνταγματικούς θεσμούς με τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, οι κάτω χώρες, η Δανία Ε, με τη Δανία ε, και είναι ε, τμήμα της ευρωπαϊκής οικογένειας και γι' αυτό πρέπει να υπάρχει μια διαφοροποιημένη προσέγγιση, μια ειδική προσέγγιση και το σύνολο των περιοχών αυτών όπως και το σύνολο των εκπροσώπων εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να ταχθούν υπέρ ενός εργαλείου ειδικού χρηματοδότησης, ειδικής χρηματοδότησης για γιατί αυτό θα έδινε τη δυνατότητα να μειώσει να μειωθεί το κακό ποσοστό αξιοποίησης κονδυλίων από τις υπερπόντιες αυτές χώρες και εδάφη. Ε, τέλος, το μέλλον του κοτονού τεράστιο θέμα. Θα ήθελα μόνο να επιμείνω σε ένα ζήτημα, το είχα πει και στην προηγούμενη συνεδρίαση. Όταν μιλάμε για τις χώρες ΑΚΕ, ξεχνάμε αρκετά συχνά ότι πάνω από το 80% των χωρών ΑΚΕ είναι μικρές νησιωτικές χώρες ε, υπό ανάπτυξη. Υπάρχουν βέβαια και μεγάλες χώρες της Αφρικής, αλλά το 80% των χωρών ΑΚΕ και παραπάνω ίσως ε, είναι μικρές νησιωτικές χώρες υπό ανάπτυξη. Και για τις χώρες αυτές ε, οι απαντήσεις ε, είναι ή θα έπρεπε να είναι ε, πολύ διαφορετικές, εντελώς διαφορετικές. Μπορούμε να προσπαθούμε να επιτύχουμε τους στόχους πολύ πιο γρήγορα στις μικρές νησιωτικές χώρες από ό,τι στις μεγάλες χώρες και γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει στην περίοδο μετά το κοτονού να υπάρχει μια καλύτερη ε, να λαμβάνεται καλύτερα υπόψη ο νησιωτικός χαρακτήρας ε, των κάποιων περιοχών ε, και ώστε να υπάρξει και η κατάλληλη στρατηγική. Και τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα της μετανάστευσης που είναι προφανώς στο επίκεντρο των ανησυχιών. Πεποίθησή μου είναι ότι 100% της αναπτυξιακής βοήθειας ε, συμμετέχει ε, στους στόχους περιορισμού της μετανάστευσης γιατί όσο αναπτύσσονται αυτές οι χώρες τόσο λιγότερο μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα υπάρχουν ε, αναχωρήσεις από τις χώρες αυτές. Όμως ε, σε γενικές γραμμές ε, δεν μπορούμε μόνο μέσω αυτής της πολιτικής ε, να καλύψουμε αυτό το θέμα που είναι θεμελιώδες, είναι μεγάλη σημασία όταν βλέπουμε τις δημογραφικές προοπτικές μέχρι το 2100 12 δισεκατομμύρια κατοίκους θα αριθμεί η γη μας. Στην Αφρική θα ζουν πάνω από 4 δισεκατομμύρια άνθρωποι. Από το 1 δισεκατομμύριο θα πάμε στα 4, τετραπλασιασμός δηλαδή σε 100 χρόνια, δηλαδή σε μια ζωή για να το πω έτσι. Ο πληθυσμός της Νιγηρίας το 2100 θα είναι περίπου 900 εκατομμύρια, δηλαδή όσο είναι σήμερα όλος ο πληθυσμός Αφρικής. Το 2100 ο πληθυσμός της Ευρωπαϊκής Υπήρου θα είναι περίπου 600 εκατομμύρια. Πρόκειται δηλαδή για έναν ε, πληθυσμό που είτε μειώνεται είτε διατηρείται και σας δίνω όλα αυτά τα αριθμητικά στοιχεία για να σας δώσω μια ιδέα των όσων μας περιμένουν. Ε, υπάρχει και το θέμα της κλιματικής αλλαγής που λαμβάνει η χώρα. Ε, κάποια ζητήματα που έχουν σχέση με αυτό θα ε, επιδεινώσουν ακόμη περισσότερο τις ε, συνέπειες ε, τις κλιματικές σε κάποιες χώρες και αυτό θα οδηγήσει σε νέες μεταναστευτικές ροές. Δεν είναι λοιπόν μόνο η αναπτυξιακή βοήθεια όπως τη γνωρίζουμε και όπως την έχουμε προσδιορίσει ε, που θα μας επιτρέψει να απαντήσουμε, να ανταποκριθούμε στην πρόκληση αυτή ε, οι απαντήσεις βρίσκονται και αλλού για τις προκλήσεις αυτές. Ολοκληρώνοντας, έχοντας έτσι μια ευρύτερη θεώρηση της αναπτυξιακής πολιτικής, βλέπουμε ότι το σύνολο των ε, πλανητικών προκλήσεων και το σύνολο των ευρωπαϊκών προκλήσεων ε, ε, γίνεται, λαμβάνουν χώρα στην Αφρική, στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό, κλιματική αλλαγή, μεταναστευτικές προκλήσεις και, θα επιμείνω σε αυτό, ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το λάβει υπόψη στην περίοδο μετά το Κοτονού, το ζήτημα της διατήρησης έχουν φύγει συνάδελφοι από τους πράσινους. Ο κύριο Αρέγκ βέβαια είναι εδώ, αχ, συγγνώμη, λάθο έκανα. Το θέμα της βιοπικιλότητα. βρισκόμαστε ε, στην έκτη, στο έκτο κύμα ε, εξαφάνισης των ειδών. Ε, τα είδη αυτά βρίσκονται κατά κύριο λόγο στην Αφρική και νομίζω ότι μέσω της αναπτυξιακής βοήθεια μπορούμε να δράσουμε αλλά εδώ ξεφεύγουμε πάρα πολύ από τον απλό δημοσιονομικό έλεγχο. Η προθεσμία καταβολής ε, ε κατάθεσης τροπολογιών είναι 6η ε, Μαρτίου. Κατά τη συνεδρίασή μας ε, με τους κοιόδης εισηγητές θα προτείνω να χορηγήσουμε την απαλλαγή για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι όλους ιδιαίτερος που αυτή η Επιτροπή δίνει πολύ σημασία στην ε, στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης και ότι όλοι οι συνάδελφοι ενδιαφέρονται πάρα πολύ και καταβάλουν και πολλή ενέργεια για αυτό το θέμα. Κυρία Σμιτ. Ευχαριστώ αγαπητέ κύριε Σίγητα, αγαπητοί συνάδελφοι. Πρώτα πρέπει να ευχαριστήσω με το ελεκτικό συνέδριο μαζί με τον εισηγητή. Νομίζω ότι είναι πολύ ισορροπημένη έκθεση αυτή με πάρα πολλά θέματα όπως ακούσατε. Το Ταμείο Ανάπτυξης καμιά φορά θεωρείται ο συνήθις ή όταν πρόκειται για αισθίε προβλημάτων. Αυτό είναι πολύ ανησυχητικό. Το τελευταίο ταμείο έχει προϋπολογισμό 30,5 δις, ε, το ενδέκατο ταμείο και 76,88 δις τα τέσσερα ταμεία. Όλα αυτά είναι μεγάλα κονδύλια για ε, να τα διαχειρίζονται χωρίς την ε, συμμετοχή του ε, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γι' αυτό η έκθεση ελέγχου έχει τόση σημασία. Ισορροπημένη έκθεση λοιπόν όπως είπα. Προσθέτω όμως ότι ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις δαπάνες ε, χρειάζεται ξεκάθαρη γλώσσα. Έχω στους εξής τομείς επιφυλάξεις. Για τα ραλ, υπόλοιπο προσεκαθά, ε, ε, για καταπιστευματικά ταμεία, τη ε, επικεφαλής, διευθύνσεων που συνεργάζονται με διεθνείς οργανισμούς. Ε, είχα κάτι έπιες επαφές και κατάλαβα ότι έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε ακόμα. Ε, άμεση δημοσιονομική βοήθεια και οι βασική δείκτες επιδόσεων. Αυτοί όλοι είναι τομείς που ε, παρουσιάζουν κάποια προβλήματα. Δεν είχα τη χαρά να μιλήσω με τον Επίτροπο Μίμητσα στην Αρούβα. Παρ' όλα αυτά όμως αντέδρασε σε κάποια σημειώματα σχετικά με ε, εντάλματα ανάκτησης και πιστεύω ότι θα υποβάλει και άλλες διευκρινήσεις. Όλοι είμαστε ε, υπέρ της διαφάνειας και όλοι έχουμε ε, λόγο να βοηθήσουμε γι' αυτό. Το Ταμείο Ανάπτυξης καλύπτει και μεγάλη γεωγραφική περιοχή. 79 αφρικανικές χώρες, ε, χώρες ΑΚΕ και επίσης ε, και στις ε, υπερπόντιες, υπερπόντιες χώρες και εδάφη πηγαίνουν κάποια χρήματα, τα περισσότερα όμως δαπανώνται στην Αφρική περίπου 30, 30 δις ευρώ. Και Έχουμε στοιχεία και για τις υπερπόντιες χώρες και εδάφη. Βέβαια εσείς ε, εστιάζετε υπερβολικά και το καταλαβαίνω στις ε, υπερπόντιες χώρες και εδάφη. Αλλά σε μια έκθεση ελέγχου ε, δεν πρέπει να τονίζουμε ιδιαίτερα τα προβλήματα των υπερποντίων χωρών και εδαφών. Λοιπόν, η έκθεση είναι επιτυχής, παρόλα αυτά όμως ε, επιφυλάσσομαι να καταθέσω πολλές τροπολογίες με διαφοροποίησεις που θεωρώ ότι χρειάζονται. Θα συνεχίσω στα αγγλικά, ακούσαμε γερμανικά και γαλλικά, έχω γράψει τις σημειώσεις μου στα αγγλικά. Λοιπόν, καταρχάς να ευχαριστήσω το ελεκτικό συνέδριο αλλά και τον εισηγητή μας τον κύριο Ματζή για την εξαιρετική του εργασία. Όπως κυρία Σμιτ θεωρώ ότι είναι επικοδομητική αυτή η έκθεση. Η πολιτική μου ομάδα λυπάται που έχουμε μειωμένε πιστώσεις για το 2015 εξαιτίας της στάση Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτό ουσιαστικά επιδίνωσε την αναπτυξιακή βοήθεια προς τις χώρες με τις οποίες συνεργαζόμαστε. 408 εκατομμύρια ευρώ το 2016 και 1 εκατομμύριο ευρώ ε, καθυστερούμενος στόκος. Επίσης, οι δαπάνες για το 2015 ε, περιέχουν ακόμα τα ε, πόρους από το 8ο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, το οποίο για 19,59. Επίσης, είναι πάρα πολύ σημαντικό να αυξηθεί η δυνατότητα λογοδοσίας, δημοκρατικού ελέγχου και να έχουμε περισσότερη διαφάνεια και μια μεγαλύτερη ορατότητα για τη χρήση των κονδυλίων αυτών και κατά αυτόν τον τρόπο θα μειωθούν επίσης και τα τέλη συναλλαγών καθώς επίσης και τα τέλη που έχουν να κάνουν με την υποβολή εκθέσεων. Θα υπάρχει ένας κοινός, μια κοινή δέσμη κανόνων, διοικητικών. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξη και τα διάφορα τέτοια ταμεία ουσιαστικά αντιμετωπίζουν τα βαθύτερα αίτια τη προσφυγική και μεταναστευτική κρίση. Τα Ευρωπαϊκά Ταμεία λοιπόν Ανάπτυξη δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για άλλου λόγου πέρα από αυτού προβλέπονται στι βασικέ διατάξει, όπω για παράδειγμα έλεγχο των εξωτερικών συνόρων και αποτελεσματική επιστροφή. Οι συνέργειες αυτή τη στιγμή ανάμεσα στον κοινοτικό προπολογισμό, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης και οι διμερείς επίσης συνεργασίες θα πρέπει να συνδυάζονται με τον κατάλληλο τρόπο προκειμένου να έχουμε πρόληψη περαιτέρω της μετασταυτικής κρίσης. Θα πρέπει επίσης να δούμε πώς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων μπορεί να συμβάλλει και αυτό με τη σειρά του, προκειμένου να έχουμε πλήρη λογοδοσία και εμπλοκή του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς επίσης και υποβολή εκθέσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συμφωνώ με τον ε, εισηγητή ότι ο κατακαιρματισμός των εργαλείων που έχουμε εδώ πέρα με ξεχωριστούς στόχους το καθένα και χωρίς μεταξύ αυτών διασύνδεση δεν επιτρέπει στο Κοινοβούλιο να παρακολουθήσει καλύτερα πώς δαπανώνται αυτά τα κονδύλια. Και κατά αυτόν τον τρόπο δεν καταφέρνουμε να κατανείμουμε τις ευθύνες και να δούμε τελικά τα κονδύλια αυτά όντως χρηματοδοτούν την εξωτερική δράση για τη μετανάστευση. Πρέπει επίσης οι δείκτες επιδόσεων να είναι σαφείς και θα πρέπει να υπάρχει λογοδοσία και στην πτυχή των δαπανών. Θα πρέπει να αποφύγουμε τον κίνδυνο λανθασμένης χρησιμοποίησης των κονδυλίων αυτών ή επικαλύψεων όσον αφορά τη χρήση των ταμείων αυτών και θα πρέπει να αποφύγουμε τα ταμεία αυτά να υποστηρίζουν τους λανθασμένους δικαιούχους. Θα πρέπει επίσης να βελτιώσουμε τη διαχείριση των ταμείων αυτών προκειμένου να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και νέα εργαλεία αντιμετώπισης κρίσεων, για παράδειγμα μέσω συνδυασμένων μηχανισμών χρηματοδότησης σε συνεργασία και με άλλους διεθνείς οργανισμούς απευθυνόμενοι σε χώρε ε, οι οποίε μπορεί να είναι δικαιούχοι πολλών διαφορετικών εργαλείων. Η αιρεσιμότητα. Ε, ναι, είμαστε υπέρ τη αιρεσιμότητα, αρκεί και εδώ πέρα να έχουμε αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα. Είμαστε υπέρ του ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ενσωματώσει το ζήτημα του κινδύνου στη διαχείριση των εξωτερικών δράσεών τη. Και εδώ πέρα βλέπουμε ότι έχουμε ένα πολύ έθραυστο περιβάλλον όπου ελοχεύουν πολύ διαφορετικοί κίνδυνοι. Οι χώρες εταίροι βρίσκονται σε διαφορετικό επίπεδο ανάπτυξης, έχουν διαφορετικές συνθήκες διακυβέρνησης. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε καλύτερη παρακολούθηση των κινδύνων αυτών. Αναγνωρίζουμε επίσης ότι μέσω της συνεργασίας αυτής, της συνεργασίας που έχουμε με διεθνείς οργανισμούς μπορούμε να αποφεληθούμε όλοι. Θα πρέπει όμως εδώ να διορθώσουμε τις αυναμίες και τα λάθη που έχουν προκύψει και να βελτιώσουμε την προβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κονδύλια από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξη θα πρέπει να γίνονται πιο αισθητά, να γίνονται πιο κατανοητά από τους Ευρωπαίους πολίτες. Επίσης, είναι σημαντικό να δούμε τι γίνεται με, με τις υπερπόντιες χώρες και εδάφη. Δεν καλύπτονται εδώ τα όσα λέγονται από το πεδίο εφαρμογή του Ταμείου αυτού και βλέπουμε επίσης ότι δεν αποτελούν τμήμα της διαδικασία απαλλαγής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να αυξήσει τις δραστηριότητες δέουσας επιμέλειας, προκειμένου όντως να διασφαλίζεται ότι τα κονδύλια αυτά φτάνουν στους τελικούς δικαιούχους και ότι δεν χάνονται τελικά ή δεν αποτελούν αντικείμενο διασπάθησης από διαμεσολαβητές. Να τονίσουμε για άλλη μια φορά ότι θα πρέπει να έχουμε ένα συγκεκριμένο αυστηρό κατάλογο κριτηρίων για την ε, επιλογή διαμεσολαβητών. Όταν γίνεται αυτό, με συνεργασία με τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προσβλέπουμε και σε μελλοντικές συζητήσεις. Αυτά είχα να σας πω για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Δεν ε, έχω άλλον στον κατάλογο. Η Κομισιόν. Γενική Διεύθυνση Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή που πρότεινε να χορηγηθεί η απαλλαγή για τα Ευρωπαϊκά ανάπτυξη 8 1 9ο, 10ο, 11ο και 11 ε, Είναι ένα έγγραφο αρκετά εξισορροπημένο που λαμβάνει υπόψη την συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά αναφέρεται και σε κάποιες αδυναμίες, ε, τονίζει τρόπους βελτίωσης, ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνει ό,τι μπορεί για να ικανοποιήσει τα αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πολλά ζητήματα πραγματεύεται αυτό το έγγραφο, δεν θα απαντήσω σε όλα. Θα ήθελα να αναφερθώ ε, στα πιο σημαντικά. Υπήρξε ένα ερώτημα για την ανάκτηση, αλλά μπορούμε ενδεχομένως να απαντήσουμε γραπτός, ε, ε, αν θέλει να μας απευθύνει και γραπτός η κυρία Σμιτ έχουν γίνει διορθώσεις, ε, ε, ε όμως ε, πολλές φορές οι ανακτήσεις δεν γίνονται γιατί ήταν, είτε δεν ήταν σωστές οι ημερομηνίες είτε δεν ήταν τα ποσά σωστά ε, πάντως υπάρχουν τα απαραίτητη αιτιολόγηση από τους ε, ε, υπεύθυνους λογιστικού ελέγχου. Όσον αφορά τον έλεγχο εξάντε, υπάρχει ένα ποσοστό σφάλματος 3,8% που είναι σχετικά σταθερό. Υπήρξε μία μικρή αλλαγή λόγω της αλλαγής της μεθοδολογίας του ελεγκτικού συνεδρίου πριν από τρία χρόνια. Είναι κάτι το πάρα πολύ δύσκολο εγχείρημα όμως ε, σε χώρες όπου υπάρχει μεγάλη αστάθεια, ε, ζώνες ένοπλων σειράξεων, εμπόλεμες περιοχές. Ε, σε γενικές γραμμές πάντως πέφτει το ποσοστό, μειώνεται ήταν το 2015 2,2%. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του ε, ποσοστού υπολείποντος φάλματος. Είναι ένα ποσοστό το οποίο ε, προκύπτει όταν έχουν γίνει όλοι οι έλεγχοι, όταν έχουν κλείσει όλες οι συμβάσεις. Ε, το ελεγκτικό συνέδριο υπολογίζει το ποσοστό ε, βάση μια συγκεκριμένης ε, χρονικής στιγμής μιας συναλλαγή. Μετά, οι διάφοροι χειριστέ ενός ε, project μπορούν να, να διορθώσουν τα ποσοστά και να κοινοποιήσουν τα αποτελέσματα του ελέγχου στο ελεγκτικό συνέδριο. Μερικές φορές όμως υπάρχει έλλειψη τεκμηρίωσης, γιατί Μιλάμε για χώρες οποίες ε, είναι αρκετά ευάλωτες και ε, η κοινωνία των πολιτών ε, δεν έχει το σύνολο των μέσων να διατηρήσει ποιοτικά αρχεία και μερικές φορές υπάρχει και μη σεβασμός των συμβάσεων. Δεν λέω ότι υπάρχει κατάφορη παραβίαση. Απλώς μερικές φορές η, σύναψη των ε, συμβάσεων ε, αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα όσον αφορά την ερεσιμότητα και το κριτήριο ε, ανάθεσης των συμβάσεων έργου. Έχουμε λοιπόν ένα σύστημα αξιολόγησης εκ των πολύ, εκ των προτέρων, πολύ προχωρημένο έχουμε μειώσει το ποσοστό ε, ε, σφάλματος, ε, τουλάχιστον του υπολοιπόμενου σφάλματος όπως εξήγησα προηγουμένως και υπάρχει επίσης και το κόστος του ελέγχου. Υπάρχει μία μείωση του κόστους αυτού του διοικητικού άχθους δηλαδή, όλα αυτά πρέπει να τα βάλουμε σε μία προοπτική. Μειώνεται το ποσοστό σφάλματος με ποσοστό κόστους ελέγχου επίσης που μειώνεται. Ε, γίνεται εκ των προτέρων έλεγχος όλων των συναλλαγών ε, μέσω των χωρών εταίρων ε, βάσει των, της σύναψης συμβάσεων έργου που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν το κάνουν αυτό οι εταίροι από μόνοι τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επί τη βάση των, ετα... των ετοιμάτων των χωρών αυτών κάνει τον έλεγχο. Βρισκόμαστε λοιπόν σε ένα σύστημα διαχείριση έμεση, το οποίο ελέγχεται πάρα πολύ λεπτομερώς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πρέπει να λάβετε υπόψη το κόστος κάθε φορά που θέλουμε να μιλήσουμε για αύξηση μείωση του κόστου ε, σφάλματος, του ποσοστού σφάλματος. Όσον αφορά τι επιδόσει τώρα, ε, το οποίο επίση αναφέρθηκε, για τα σχέδια που μπλοκάρουν, που δεν προχωρούν και που θεωρούνται κόκκινα, χαρακτηρίζονται κόκκινα. Εμείς κάνουμε μια παρακολούθηση πολύ στενή ε, ε, με πρώτερο αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βάσει του άρθρου 16 ε, δίνουμε τη δυνατότητα από τη μία χρονιά ε, στην άλλη ε, να εξελιχθούν τα προγράμματα. Εντοπίζουμε τα βασικά ζητήματα που είναι τα ζητήματα υποδομής, διαχείρισης από τα κράτη, εταίρους κλπ. Και αξιολογούμε τα διορθωτικά μέτρα που ελήφθησαν. Τώρα, ε, πολλές φορές πρόκειται για έγγραφα, για προγράμματα που είναι κόκκινα ή πορτοκαλί ε, και τα οποία θεωρούμε ότι μπορούν να κλείσουν γιατί ούτως ή άλλως δεν επιτυγχάνουν τους στόχους τους. Ε, επί 55 προγραμμάτων το 2015, 100 46 ε, ε, ε, βελτιώθηκαν, ε, ε, όμως δυστυχώς υπάρχουν άλλα τα οποία χαρακτηρίζονται μετά κόκκινα ε, για διάφορους λόγους. Ένα ακόμη ε, σχόλιο για να μην υπάρχει παρεξήγηση. Καταλαβαίνω να μιλούμε για δραστηριότητα εξωτερική, εξωτερικούς εταίρους όταν μιλάμε για διεθνείς οργανισμούς ε, ή για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ε, ο οργανισμοί που πρέπει και εκείνοι να συνεισφέρουν στην εφαρμογή της ε, αναπτυξιακής πολιτικής της Ένωσης και που πρέπει επίσης να ελέγχονται και συμφωνούμε απολύτως με τις προτάσεις που έχει υποβάλει ο εισηγητής επί των σημείων αυτών. Ε, θα ήθελα πέρα από την διαφάνεια Συμφωνούμε και από αυτού ε, ότι δεν πρέπει να υπάρχει κατακαιρματισμός των μέσων. Ε, θέλουμε να συμμετέχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην εποπτεία. Ε, έχουμε καλέσει μάλιστα σε διάφορες διαχειριστικές επιτροπές να συμμετέχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Ε, συμφωνούμε λοιπόν απολύτως ε, ε, ε με αυτά. Ε, ο έλεγχο γίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να σα πω για παράδειγμα, η δήλωση αξιοπιστία για το Γενικό Διευθυντή τη ΔΕΦΚΟ. Θα κάνει μια δήλωση αξιοπιστία στο σύνολο και για, την και για το Ταμείο Ανάπτυξη και τα καταπιστεύματα και τα ταμεία τα οποία γυρίζονται τα κράτη-μέλη. Τα trust fund όμως θα είναι σε διαφορετικές ομάδες ε, ως προς τη δήλωση αξιοπιστία. Είτε πρόκειται για τον ε, λογιστικό έλεγχο, για την διεθνή συνεργασία και ανάπτυξη, είτε πρόκειται για την, αλυσί, για την ε, αλληλουχία των εκθέσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της δήλωσης αξιοπιστίας μέχρι το Γενικό Διευθυντή, είτε για την ε, μελέτη, τις μελέτες ε, ε, για το ποσοστό υπολοιπόμενου σφάλματος. Και θα ολοκληρώσω λέγοντας, επειδή ετέθηκε το ζήτημα για το African Peace Facility, Υπάρχει ένα σχέδιο δράση το οποίο έχουμε δρομολογήσει. Όπω είπατε, οι εσωτερικέ υπηρεσίε λογιστικού ελέγχου, επειδή του ζητήσαμε, ε, επειδή είχαμε δεσμευθεί να ε, ασχοληθούμε με την εφαρμογή γενικότερα, μα είπε λοιπόν η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου ότι τα περισσότερα μέτρα έχουν εφαρμοστεί. Τούτου λεχθέντος βέβαια, εξακολουθούμε να θεωρούμε σήμερα ότι η Αφρικανική Ένωση δεν είναι σε θέση να περάσει το pillar assessment, οπότε εμείς δεν θέλουμε να άρουμε την επιφύλαξη για το Peace Facility και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τις ε, συναλλαγές πολύ πολύ προσεκτικά. Κάτι ακόμη. Ο έλεγχο που γίνεται από την Εσωτερική Υπηρεσία Ελέγχου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, δεν τοποθετείται επί τη παρατυπία, επί των παρατυπιών των συναλλαγών. Δεν υπάρχουν παρατυπίε ως προς τα μη επιλέξιμα ε, ταμεία. Ε, ο κίνδυνος αφορά πάντα έναν, έναν πιθανό κίνδυνο. Από το 2009 ε, είχαμε υπογράψει ένα μνημόνιο κατανόησης με την Αφρικανική Ένωση ε, με την Αφρικανική Ένωση είχαμε ζητήσει κάποια περισσότερα πράγματα αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσε να τα καλύψει η Αφρικανική Ένωση και από το 2015 και μετά ε, παρακολουθούμε το ε, ε, σύστημα εκ του σύνεγγυς. Θα σταματήσω εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την γνωμοδότηση. Λοιπόν, τελειώσαμε στο σημείο αυτό της ημερήσιας διάταξης και της ανοιχτής συνεδρίασης. Η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών 6 Μαρτίου 2017, 2 το απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζομαι με τους συντονιστές που παρακαλώ να μείνουν στην αίθουσα. Οι υπόλοιποι παρακαλώ να εγκαταλείψουν την αίθουσα το ταχύτερο δυνατόν. Λύεται η συνεδρίαση.